Καλημέρα σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ε, πρώτα απ' όλα βέβαια θα καλωσορίσουμε τον νέο Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, τον ε, Υπουργό Γεωργίας της ε, Λιθουανίας, ε, τον κύριο Βιρτζίλιους Γιούκνα. Αγαπητέ Βιρτζίλιους, αναλαμβάνεις την Προεδρία σε μια καθοριστική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Γεωργία και όπως πολύ καλά γνωρίζεις ε, περάσαμε μία περίοδο ε, σε βάθος διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής υπό την Ιρλανδική Προεδρία. Στις 26 Ιουνίου του περασμένου έτους καταλήξαμε σε μία πολιτική συμφωνία που αφορά στο μεγαλύτερο μέρος ε, των θεμάτων που έχουν σχέση με τους τέσσερις φακέλους μεταρρύθμισης της κοινή αγροτικής πολιτικής. Τώρα λοιπόν, αγαπητέ Πρόεδρε, υπό τη Λιθουανική Προεδρία καλούμεθα να δώσουμε τελική μορφή σε αυτή τη μεταρρύθμιση και ελπίζουμε το συντομότερο δυνατόν να καταλήξουμε όσον αφορά στις ε, εκκρεμούσες υποθέσεις. Είχαμε μια συζήτηση εχθές ε, με τους ε, συντονιστές, τους συζητητές και τους σκιώδης για τα θέματα τα οποία έχουν ακόμα εκκρεμότητες και είμαστε πεπισμένοι ότι υπό τη δική σου την καθοδήγηση θα μπορέσουμε ταχύτατα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και για τα θέματα αυτά. Και αυτό για να κατορθώσουμε να ε, μπορέσουμε να κλείσουμε όλους τους ε, φακέλους της κοινή ε, αγροτικής πολιτικής και με τον τρόπο αυτό να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην ε, Επιτροπή Γεωργίας και στην Ολομέλεια. Σου εύχομαι λοιπόν σε σένα Βιτζίλιους και στην Λιθουανική Προεδρία να ευοδοθούν οι προσπάθειές σου, όχι μόνο για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά και για ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητήσαμε χθε με τον κύριο Ντές, σχετικά με τα ε, μεταβατικά μέτρα. Εύχομαι λοιπόν να καταστεί δυνατόν να υπάρξει πρόοδος και σε άλλα ε, νομοθετικής φύσεως θέματα κυρίως ε, όσον αφορά την προστασία των φυτών και των ζώων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα και προσβλέπουμε πρόοδο κατά τη διάρκεια της ε, Λιθουανικής ε, Προεδρίας. Σε ευχαριστώ λοιπόν που ήρθες και θα σου δώσω τώρα το λόγο για να μας παρουσιάσεις το πρόγραμμα της Λιθουανικής Προεδρίας. Και μετά, ως συνήθως, θα δώσω το λόγο στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και μετά μπορεί να παρέμβει όποιος επιθυμεί για να υποβάλει ερωτήσεις στο νέο πρόεδρο. Πρόεδρο. Αγαπητέ Βιτζίλη, έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πάρα. αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίε και κύριοι. Η Λιθουανία για πρώτη φορά στην ιστορία της αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μεγάλη μου τιμή, επομένως. Να είμαι ο Προεδρεύων του Συμβουλίου και να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Προεδρίας μας, γιατί πρόκειται για μια ιστορική πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να έχουμε τα ενία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τώρα που η Κροατία έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε 28 τα κρατημέλη. Επίσης, πρόκειται και για μια ευκαιρία. Ευκαιρία να δείξουμε ότι μια μικρή χώρα είναι θέση να λύσει προβλήματα με τρόπο αποτελεσματικό. Sieksime sažiningai dalyvauti teisėkuros ir sprendimų Πρόκειται για μια ευθύνη. Αυτή η ευθύνη μας γεμίζει με ικανοποίηση όμως και θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε έτσι με έναν τρόπο έντιμο να διαχειριστούμε την διαδικασία λήψη αποφάσεων και έτσι να εξασφαλίσουμε την συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορέσουμε επίσης να εμπλέξουμε ε, όλους όσους πρέπει σε αυτή τη λήψη αποφάσεων από την άλλη μεριά όμως ε, ξέρετε ότι ως Πρόεδρο του Συμβουλίου θα, θα πρέπει να συνεργαστώ μαζί σας που είστε εταίροι μας, που είστε συνομοθέτες και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους συμπολίτε μας. Οπότε και εγώ θεωρώ ότι θα συνεργαστούμε και επίσης πρόκειται όλα αυτά τα θέματα που έχουμε δεκπεριώσουμε ε, να τα αναλάβουμε από κοινού. Πρώτα πρώτα. Να σας πω ποιες είναι οι προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας. Το πρόγραμμα της Προεδρίας θα εστιαστεί ίσως να έχουμε μια αξιόπιστη ανοιχτή Ευρώπη με ανάπτυξη. Θα είναι σφαιρικό πρόγραμμα. Πρόκειται να καλύψουμε την δημοσιονομική σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Ιδίω την απασχόληση των νέων. Ιδίω όσον αφορά την ε, ενία αγορά, αλλά επίση θα έχουμε και του στόχου που σχετίζονται με την ε, ασφάλεια. Ως φόδος του Συμβουλίου Αλίας και Γεωργίας θα μπορέσω να προωθήσω κάποιες πολιτικές οι οποίες θα είναι φιλικές στο περιβάλλον, θα είναι καινοτόμε και θα μπορέσουμε γενικά να εξελίξουμε ε, τον τομέα τον αγροδιατροφικό αλλά και τον αλληλευτικό. Τώρα να σας πω ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την γεωργία. Πρώτα πρώτα, να ολοκληρώσουμε την μεταρρύθμιση της κοινή ερωτικής πολιτικής. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά, διότι ολοκληρώσαμε τη δέσμη μέτρων για την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ κατόπιν διαπραγματεύσεων. Είχαμε ε, συζητήσεις, έντονες πάνω από 40 τριμερείς διαλόγους και πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα προς μίμηση. Ότι δηλαδή τα τρία θεσμικά όργανα είναι στέση να συμφωνήσουν σε ζητήματα ε, υψής πολιτικής σημασίας τώρα μέσα στο θεσμικό περιβάλλον της συνθήκης της Λισαβόνας. Επίσης και προσωπικά θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε, αλλά και τους ηγητές, τον κύριο Λουίς Καπουλασάντος και τον κύριο Μισελ Ντοντέ, αλλά και τον κύριο Τζοβάνι Λαβία και άλλα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, διότι συνέβαλαν εις το να πετύχουμε μια συμφωνία για αυτό μας τον κοινό στόχο. Η βιώσιμη και αποτελεσματική κοινή ερωτική πολιτική. Επίσης, θα πρέπει να ευχαριστήσω και τον προκατοχό μου, τον κύριο Σάιμον Κόβενι, αλλά και τον Επίτροπο Τσόλος, διότι επιτέλεσαν εξαίρετο έργο και βοήθησαν στο να συμφωνήσουμε με την Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου. Ένα επίτευγμα πάρα πολύ αξιόλογο, το οποίο αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, πολλά μπορούμε να καταφέρουμε. Οπότε, Μετά από αυτή την ε, διοργανική πολιτική συμφωνία για τη δέσμη μέτρων της μεταρρυθμιστής ΚΑΠ, η Προεδρία τώρα έχει ως στόχο να ολοκληρώσει την προσπάθεια η οποία σχετίζεται με την έγκριση και έγκαιρη θέση σε ισχύ αυτή της δέσμη μέτρων για την ε, καινούργια κοινωνική πολιτική. Επομένως, έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά και δύσκολη. Σας βεβαίω συνάδελφε ότι όλα όσα συμφωνήθηκαν στο Λουξεμβούργο, τις Βρυξέλλες και το Στασβούργο ε, τις τελευταίες 15 μέρες πρόκειται να αποτυπώνονται στα τελικά σχέδια κειμένου. Επίσης, πρόκειται στιάσουν την προσοχή μας στο να συζητηθεί και να εγκριθεί μια πρόταση για τους αναγκαίους μεταβατικούς κανόνες για κάποια σημεία της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, ιδίως όσον αφορά τις ε, άμεσες πληρωμές, άμεσες καταβολές και επίσης την ανάπτυξη της υπαίθρου. Όπως γνωρίζετε, με αυτές τις προτάσεις θέλουμε να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση από τα όσα σήμερα ισχύουν σε όσα θα διέπουν την καινούργια την ευρωτική πολιτική μετά τη μεταρρύθμιση. Θα πρέπει ε, αυτού του είδους οι μεταβατικοί κανόνες θα πρέπει να εγκριθούν και να εφαρμοστούν το 2014. Οπότε και η Λιθουανική Προεδρία πρόκειται να επιδιώξει συμφωνία και στο Συμβούλιο αλλά και σε ε, διοργανικό επίπεδο. Πρόκειται για μια κοινή πρόκληση και κοινή ευθύνη. Να μπορέσουμε να έχουμε ξεκάθαρους κανόνες και να παράσχουμε στους ε, γεωργούς τις οικονομικές εγγύησεις για αυτήν την μεταβατική περίοδο. Επίση, τώρα θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Αλμπερντέ, ο οποίο είναι ο συγητή αυτή τη σημαντική έκθεση. σε συνάδελφοι θα πρέπει από κενού να ενεργήσουμε συντονισμένα αλλά και γρήγορα. Πάολο, αγαπητέ πρόεδρε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πρόκειται να συνεργαστούμε με τρόπο θετικό και αποθετικό με την Επιτροπή σα ακριβώ όπω έγινε και στο παρελθόν. Και τώρα να στραφούμε στι υπόλοιπε προτεραιότητε του προγράμματο τη Προεδρία. πρώτο, πρώτα. Κάνουμε τον των ζώων, υγεία των ζώων, ε, τα φυτογειονομικά, καθώς υπήρχαν και τα σχετικά με τις ε, ζωοτροφές και τα είδη διατροφής. Έχουμε ε, αυτή τη δέσμη των πέντε προτάσεων όσον αφορά αυτά τα ζητήματα για ούτως ώστε να μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα νομικό πλαίσιο. Στις 6 Πέμπτου, ενεστώτος έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε δημοσιότητα αυτή την ε, δέσμη των πέντε μέτρων των πέντε προτάσεων, ούτως ώστε να έχουμε ε, εφαρμογή των προτύπων που ισχύουν για όλη την διατροφική αλυσίδα. Η Προεδρία θα επιδιώξει την πρόοδο σε αυτά τα ζητήματα πιο συγκεκριμένα για τον νέο κανονισμό για την υγεία των ζώων για την ε, πρόταση που θα αφορά τον κανονισμό ε, για τα φυτογειονομικά για το αναπαραγωγικό υλικό, την παραγωγή του για τη θέση του σε εμπορία, αλλά επίσης και για τους επίσημους ελέγχους της διατροφικής αλυσίδας. Το σχέδιο κανονισμού τώρα, όσον αφορά τη διαχείριση του πλαισίου για τις δαπάνες της περίοδου 2014-2020 όσον αφορά τη διατροφική αλυσίδα, τα ε, ιατρικά και τα φυτογενομικά πρόκειται να μας εξασφαλίσει μια ομαλή ροή των πόρων όσον αφορά τα προγράμματα τα οποία θα τρέξουν τα κρατημέλη. Επίσης, αυτό θα, όφερα, θα αφορά και την αντιμετώπιση των επιδημιών επιζωδιών Πρόκειται για αυτού του κανονισμού. Επομένω, οι οποίοι πρόκειται να εγκριθούν και θα τεθούν σε ισχύ από το 2014 και μετά και γι' αυτό και εμεί πρόκειται ιδιαίτερω να προσέξουμε την ανάλυση αυτή τη πρόταση, να καταλήγουμε σε πολιτική συμφωνία περί τα τέλη τη Προεδρία μα. Κύριε Πρόεδρε, εξόπινοι κύριε βουλευτέ, κυρία Λεμπρά, που είστε η εισηγήτρια, ε, υπολογίζουμε και στην δική σα συνεργασία. Και σας διαβεβαιώ ότι επί τη βάση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Λιθουανία επίσης είναι έτοιμη να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις ούτως ώστε να έχουμε πρόοδο και στην αναθεώρηση των ε, φαρμάκων ε, την κτηνιατρική τις οδηγίες ε, τις σχετικές με τις τροφές που χορηγούνται στα ζώα στα πλαίσια της ε, κτηνιατρικής φροντίδας και τα ε, ζωοτεχνικά. Τώρα για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά το πώς θα προωθήσουμε κάποια μέτρα για τις ε, εξαγωγές. Θα αρχίσουμε τις επαφές για το σχέδιο κανονισμού όσον αφορά ε, την ενημέρωση, τις πληροφορίες και κάποια άλλα μέτρα για προώθηση αγροτικών προϊόντων, τόσο ώστε να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο και σε αυτό το μέτωπο. Ο προγευευτικά τώρα. Πρόκειται για ένα τομέα πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια της ε, Γεωργίας. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε κι άλλο τη θέση του παραγωγού και των νομικών προσώπων που τους εκπροσωπούν, αλλά και την ε, διαπραγματευτική τους ισχύ. Οπότε και θέλουμε να εξετάσουμε τι δέσμη μέτρων που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει σχέδιο κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά τα προκυπευτικά. Επίσης, θέλουμε να καλύψουμε την ε, οργάνωση της κοινή ε, οργάνωσης αγοράς στα προκυπευτικά η Λιθουανική Προεδρία πρόκειται να προωθήσει βιώσιμη δασοπονία στα κρατημέλη. Και πρόκειται στο Συμβούλιο να συζητήσουμε και να εγκρίνουμε κάποια συμπεράσματα για τη νέα στρατηγική για τα δάση νέο μέσο πολιτικής δασομονίας, το οποίο θα στηρίζεται στην επικουρικότητα ε, και στον σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων. Επίσης θα προσέξουμε το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όσον αφορά τώρα την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας ω προς τη συνθήκη της Λισαβόνας είμαστε αποφασισμένοι σε συνεργασία μαζί σας να συνεχίσουμε την ε, πορεία της ευθυγράμμισης της υπόλοιπης ε, διατροφική και γεωργική νομοθεσία με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Με χαρά μου πρέπει να σας αναφέρω ότι περί τα τέλη Ιουνίου δόθηκε το πράσινο φως όσον αφορά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις που αφορούσαν κάποιες διαπραγματεύσεις για εμπορικά προϊόντα. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί βουλευτέ, πρόκειται για μια σύντομη παρουσίαση των βασικών προτεραιοτήτων τη ε, Προεδρία μα όσον αφορά το γεωργικό τομέα. Και όπω διαπιστώνετε, πρόκειται να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα κατά το επόμενο εξάμεινο. Μας περιμένει πολλή δουλειά και γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε τρόπο αποτελεσματικό και δυναμικό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα την Επιτροπή σας για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε. Με μεγάλη μου χαρά. Διαπιστώνω ότι οι προκάτοχοι έχουν προλιάνει το έδαφος για αυτήν την συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. και με σένα αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητέ Παύλο, αλλά και με άλλους ε, βουλευτές σε διάφορες συναντήσεις. Οπότε και εγώ και προσλέπω σε αυτή την πετυχημένη μας συνεργασία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την προσοχή σας κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ να απαντήσω τυχόν ερωτήσεις που έχετε εσείς ή τα μέλη της Επιτροπής. Και πάλι ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ε, σε ευχαριστούμε αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ Βιρτζίλιους. Ε, το πρόγραμμα της ε, Λιθωνικής Προεδρίας είναι πάρα πολύ φορτωμένο και γι' αυτό λοιπόν αν θέλετε μπορείτε να παρέμβετε ευθύ αμέσω. Ε, ως συνήθως θα ξεκινήσουμε με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Κατόπιν θα ακολουθήσουν οι σκιώδεις ηγητές και μετά όλοι οι άλλοι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Άλμπερτ. Έχει το λόγο Άλμπερτ. Άλμπερτ Ντε Ε, πρόεδρε ε, και Προεδρεύοντα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω αλλά είχα μία συνάντηση με μία ομάδα Βαβαρών και καθυστέρησα λιγάκι στη συνάντηση αυτή. Γνωρίζω κύριε Υπουργέ ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε έτσι ώστε το επόμενο εξάμεινο να ε, προωθήσετε με ταχύτητα την κοινή γεωργική πολιτική και τις μεταρρυθμίσεις. Επειδή σας γνωρίζω, ε, το γνωρίζω αυτό για σας, αλλά και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και έτσι ώστε όλα αυτά που είναι απαραίτητα για το 2014 να εφαρμοστούν έγκαιρα. Έχουμε μόνο το εξή πρόβλημα, ότι στην έκθεση αυτή είμαστε αναγκασμένοι πολλά να τα συμπεριλάβουμε σε παρένθεση, να είναι σε κρεμότητα, γιατί πάρα πολλά εξαρτώνται άμεσα από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και μόνο όταν ολοκληρωθεί αυτό θα μπορούμε να καταλήξουμε κι εμείς. Σας ε, υπόσχομαι λοιπόν ότι θα είμαι σε πολύ στενή επαφή μαζί σας ε, για να προχωρήσουμε σε πράξεις. Σας συγχαίρω επίσης για το πρόγραμμα που παρουσιάσατε. Πραγματικά είναι πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα αυτό και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα τα προωθήσετε όλα με μεγάλη ταχύτητα. Ε, το πόσο επιτυχώς εργάζεται μια Προεδρία, αυτό δεν έχει άμεση συνάρτηση με το μέγεθος της χώρας, γιατί διαπιστώσαμε ότι ειδικά οι μικρές χώρες προσπαθούν ε, πάρα πολύ να σημειώσουν ε, επιτυχημένη Προεδρία εγώ έχω πάει επανειλημμένα στις χώρες της Βαλτικής, αυτοχαρακτηρίζομαι φίλος των χωρών της Βαλτικής και είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι θα τα καταφέρετε πάρα πολύ καλά. Επίσης το ΕΛΚ το επόμενο εξάμεινο δεν θα φυστεί κόπου και χρόνου έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και είμαι στη διάθεσή σας, ανά πάσα και στιγμή μπορώ να είμαι σας. Ο κύριος Κάπουλα Σάντος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ξεκινήσω καλωσορίζοντας τον νέο προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για η Λιθουανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε όλοι ίσοι. Δεν υπάρχουν μεγάλες και μικρές χώρες. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι η Λιθουανία θα ασκήσει με εξαιρετικό τρόπο την Προεδρία της και θα είμαι πραγματικά στο πλευρό σας για να συνεισφέρω και εγώ σε αυτήν την επιτυχία. Με μεγάλη προσοχή άκουσα την παρουσίαση του προγραμματός σας. Η νομοθετική διαδικασία είναι εν εξελίξη και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε αυτό το δεύτερο εξάμεινο που πάντα είναι λίγο συντομότερο από το πρώτο όσον αφορά τις εργάσιμες ημέρες να είναι αποτελεσματικό. Όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές και την ανάπτυξη της υπαίθρου Υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να τα επεξεργαστούμε. Κύριε Υπουργέ, το Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά έχει δείξει αδιαλαξία. Έχουμε παραμείνει σταθεροί στη θέση μας και είμαστε αρμόδια αρχή νομοθετική Ξέρετε όμως ότι η θέση μας έχει σήμερα ενισχυθεί. Η Προεδρία της ε, Ιρλανδίας αρχικά είχε πει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συζητηθεί το θέμα σε αυτό το επίπεδο, θα πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο Συμβουλίου. Τελικά όμως είδαμε ότι το θέμα επανήλθε σε μας, θα πρέπει λοιπόν να συναποφασίσουμε ιδιαίτερα για αυτά τα πέντε θέματα τα οποία παραμένουν εκρεμή. Κύριε Υπουργέ, τι περιθώριο ελιγμού και διαπραγμάτευσης έχετε και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρω εδώ την ενίσχυση των θέσεων του Συμβουλίου. Ο Υπουργός Κόβενη παρουσίαζε θέσεις οι οποίες φυσικά δεν ήταν δικές του, ήταν θέσεις του Συμβουλίου. Ήσασταν παρόν κύριε Υπουργέ. Ελπίζουμε λοιπόν να αλλάξει η θέση του Συμβουλίου, γιατί αν δεν αλλάξει, εάν ακούσουμε ότι ήδη έχει αποφασιστεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε Υπουργέ, τι περιθώριο διαπραγμάτευσης έχετε. Εμείς έχουμε μια εντολή, είμαστε διατεθειμένοι να δείξουμε περισσότερη ευελιξία για να συμφωνήσουμε προς συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και η διαπραγμάτευση. Χρειαζόμαστε όμως ευελιξία και οι δύο πλευρές θα πρέπει να υποχωρήσουν. Μέχρι τώρα όμως υπήρχε απόλυτη αδιαλαξία από μέρους του Συμβουλίου. Κύριε Υπουργέ, σας ξαναρωτάω και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν σας λέω να μας υποβάλλετε εδώ την συμβαστική σας ε, πρόταση το Σεπτέμβριο θα υποβληθεί από εμάς, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μία συμβιβαστική πρόταση. Πείτε μας λοιπόν τι περιθώριο διαπραγμάτευσης έχετε. Εάν έχετε βεβαίως. Θα θέλαμε να ξέρουμε. Ευχαριστώ Λουίς. Ο Τζορτζ Λάιον και μετά ο κύριος Νίκολσον. Uh, thank you, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον Υπουργό. Του εύχομαι κάθε επιτυχία για τους επόμενους έξι μήνες. Βεβαίως έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε. Έχουμε το θέμα της ευημερία των ζώων, της κατεξουσιοδότησης πράξης, και βεβαίως την ε, συμφωνία για την αναθεώρηση της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής η οποία καταρχήν έχει αποφασιστεί από την Ιρλανδική Προεδρία τον Ιούνιο. Όπως είπε και ο προηγούμενος ε, ομιλητής, γνωρίζουμε την θέση του Συμβουλίου τον τελευταίο καιρό και βεβαίως υπάρχουν και τα στοιχεία του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά και η κάποια ευελιξία στον ε, τριμερή διάλογο που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Τι δυνατότητες έχετε για να υπάρξει πρόοδος και να επιτευχθεί τελικά το αποτέλεσμα που όλοι ευελπιστούμε. Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. George. Ο Τζιμ Νίκολσον. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, Υπουργό όπως το έκαναν και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι πριν από εμένα. Ε, είσαστε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος, έχετε μπροστά σας έξι πολύ σημαντικούς μήνες. Ε, κατ' ουσίαν βέβαια πέντε είναι οι μήνες αυτοί, αλλά ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά για αυτό το χρονικό διάστημα. Ε, πολλοί είπαν ότι είσαστε ένας τίμιος διαπραγματευτής ε, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι θα προσπαθήσετε πάση θυσία να ολοκληρώσετε το έργο μας. Ίσως πρέπει να πούμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται στη μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής. Κατά την άποψή μας ε, επίκειται ένα πολύ σημαντικό καθήκον γιατί Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε το εξή. Όταν φτιάχνουμε ένα σπίτι, φτιάχνουμε του τοίχου, βάζουμε τη σκεπή, αλλά για να ολοκληρωθεί το σπίτι λείπουν οι λεπτομέρειε. Και το λέμε εξάλλου, ο διάβολο κρύβεται στι λεπτομέρειε. Όπω είπε και ο Τζορτζ, ε, αναφέρθηκε στι κατεξουδότηση πράξη, στη δική μα τη συμβολή. Δεν θα εκπλήσεστε λοιπόν ότι εγώ ε, στηρίζω αυτά που είπαν και ο Λουί και ο Τζορτζ και θα ήθελα ευθέως να σας ρωτήσω και θα ήταν χρήσιμο αν μπορείτε να μας πείτε τι είδου ευελιξία και πόση ελευθερία σας έχει προσφερθεί για να χειριστείτε τα θέματα. Γιατί θέλω να σας πω ότι για μας αλλά και κυρίως για τους εισηγητές δεν υπάρχει, μας έχουν πει ότι δεν υπάρχει περιθώριο λιγμών. Κατόπιν τούτου για μας αυτό ήταν πολύ δύσκολο να το αποδεχτούμε. Κρεμούν λοιπόν πολλά θέματα, όλοι μας το γνωρίζουμε αυτό, αλλά θέλουμε να συνεργαστούμε. Και πραγματικά ελπίζω ότι ήρθατε εδώ όχι μόνο με ένα χέρι, αλλά με δύο χέρια ελεύθερα και όχι δεμένα πιστάγκονα. και θα ευχόμουν να μην σας ε, δεσμεύσουν γιατί για μας την Επιτροπή αυτή με τη συνθήκη της Λισαβόνας και τη δυνατότητα συναπόφασης έχουν ε, ανοίξει πολλές ευκαιρίες. Ίσως λοιπόν τελικά όλοι μας νιώσουμε περήφανοι αλλά μπορεί και οι δύο πλευρές να κάνουν λάθη και πρέπει να μάθουμε από όλα αυτά και οφείλουμε επίσης να συνεργαστούμε γιατί αν δεν συνεργαστούμε φοβάμαι ότι η κοινή γεωργική πολιτική και η γεωργοί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποφέρουν. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας ε, και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας. Πολύ ωραία. Ο Μάρτιν έχει το λόγο κύριε Υπουργέ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτή την ε, πρώτη προεδρία της ε, Λιτουανίας γιατί δική σας τη χώρα πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση. Αυτό που καλείστε να κάνετε είναι να ορίσετε τις ε, λεπτομέρειες της μεταρρύθμισης της ΚΑΠΑ. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά αυτό που έχει τώρα σημασία είναι να δούμε λιγάκι τις λεπτομέρειες. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά που εκκρεμούν και δεν έχουμε ακόμα κείμενα μπροστά μας για πολλά θέματα. Όσο λοιπόν δεν έχουμε συγκεκριμένα κείμενα δεν μπορούμε και να ψηφίσουμε. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι οι λεπτομέρειες και πολλές φορές οι λεπτομέρειες είναι πιο σημαντικές από το να ε, φτιάξει κανείς ένα ολόκληρο σπίτι. Συγκεκριμένο παράδειγμα είχαμε κάποιες ε, συζητήσεις ε, σχετικά με την διαμόρφωση των ε, οικολογικών εκτάσεων. Τώρα, κατά πόσον θα συμφωνήσουμε ή όχι, εξαρτάται από το κατά πόσον στις εκτάσεις αυτές θα χρησιμοποιούνται ζυζανιοκτώνα ή όχι. Αυτό το θέμα εκρεμεί. Ένα άλλο θέμα ε, το οποίο νομίζω το έθιξαν και οι προαλήσαντες, πολύ σημαντικό, είναι οι εκκρεμότητες. Οι παρενθέσεις δηλαδή που υπάρχουν στα κείμενα, ε, τελικά και αυτές να εξαφανιστούν. Και αυτό που εκκρεμεί, και αυτό έχει μεγάλη σημασία ε, με την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, το θέμα του ανώτατου ορίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο, όπως και η εξωτερική σύγκληση και η ευελιξία ανάμεσα στους πολίνε ή πυλώνες ή χραματοδοτές χρηματοδότηση, όλα αυτά δεν είναι λεπτομέρειες, είναι καθοριστικά σημεία της ε, μεταρρύθμισης. Και ξέρετε ότι εμείς ως πολιτική ομάδα δεν μπορούμε να δεχτούμε τελικά το Συμβούλιο να πει «Ξέρετε, δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε γιατί τα θέματα αυτά τα έχουν ήδη συζητήσει οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων». Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε και εδώ λοιπόν έρχεται ο δικός σας ο ρόλος ε, να πείτε ότι θα ανοίξουμε το πακέτο και στον επόμενο τριμερή διάλογο το Σεπτέμβρη θα συζητήσουμε ειλικρινά χωρίς παροπίδες για να μπορούμε να εξαντλήσουμε τα θέματα ως προς τη συζήτηση τουλάχιστον. Κατά τα άλλα, για μας βέβαια είναι σημαντικό να καθορίσουμε τη διαδικασία για το 2014. Ο κύριος Ντες ε, ανέφερε το θέμα αυτό, αντιμετωπίζουμε μεγάλη πίεση χρόνου και νομίζω ότι για το 2014 θα πρέπει να υπάρξει ε, μια ικανοποιητική ρύθμιση ε, και όλα αυτά θα πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει το Σεπτέμβρη. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση έτσι ώστε όλα αυτά να περάσουν στην μεταβατική διαδικασία και δεν είναι λίγο το να το οργανώσετε όλο αυτό. Επίσης, ευθύς εξ αρχής αναφερθήκατε σε ένα τεράστιο πακέτο που έχει κατατεθεί, δηλαδή την προστασία ε, των ζώων, των φυτών, οι σπόροι. Όλα αυτά είναι μεγάλες ε, προκλήσεις, ε, γιατί πρέπει να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά επί της ουσίας. Η δημοσιότητα, η κοινή γνώμη, έχει στρέψει την προσοχή της στο θέμα των σπόρων και εμείς πρέπει να δείξουμε μετά τη Λισαβόνα ότι αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και θα προσέξουμε για τις λεπτομέρειες. Σας εύχομαι λοιπόν για τους επόμενους μήνες ε, καλή επιτυχία και όπως σας είπα δεν θα έχετε ε, λιγότερη δουλειά από την Ιρλανδική Προεδρία και με τον τριμερή διάλογο εμείς αποδείξαμε ότι ως Κοινοβούλιο είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε ομόφωνα, να περάσουμε τη θέση μας απέναντι στο Συμβούλιο και νομίζω λοιπόν ότι από κοινού θα μπορέσουμε μαζί με το Συμβούλιο να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα μέτρα της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Ε, πρέπει να σας πω λοιπόν ότι έχετε την υποστήριξή μας ε, που ελπίζω ε, η υποστήριξη αυτή να είναι χρήσιμη και για τους επόμενους μήνες. Ευχαριστούμε πολύ. Άγνιου και μετά Ρούμπιξ. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Δεν θα μιλήσω πολύ για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, διότι βεβαίως δεν μπορείτε να εικονοποιήσετε τόσες πολλές φιλοδοξίες, τόσο πολλά επίπεδα, τόσο πολλά ε, διαφορετικά αιτήματα και πολιτιστικά επίπεδα. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι πριν από 18 μήνες δεν θα έπρεπε να υπήρχε ούτε ένα αυγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο να ε, παράγεται με βιομηχανικό τρόπο σε τυποποιημένα ορνηθοτροφία. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό συνεχίζει να ισχύει. Συνεχίζουν να παράγονται με αυτόν τον τρόπο αυγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, πώς αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς την παραγωγή και την διάθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενετικά τροποποιημένης σόγιας και γάλατος από τη σόγια, το οποίο συνεχίζει να παράγεται στην Αμερική και οι Ηνωμένε Πολιτείες επιμένουν και συνεχίζουν να τροφοδοτούν την ευρωπαϊκή αγορά με αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι γενετικά τροποποιημένα, ισχυρίζονται όμως ότι δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτός ο κίνδυνος συνεχίζει ιδιαίτερα από τη στιγμή που παρουσιάζονται κάποια προϊόντα σαν μη γενετικά τροποποιημένα και αυξάνεται η τιμή Εγώ χρησιμοποιώ αυτά τα προϊόντα και ο τόνος έχει φτάσει πια τα 600, τις 650 λίρες. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε με αυτές τις τιμές. Οι αγρότες μας μας λένε ότι δεν είναι δυνατόν πλέον να χρησιμοποιείται η σόγια με τις τιμές αυτές. Αυτό λοιπόν που θα είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να αυξάνονται οι εισαγωγές α, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της τεράστιας διαφοράς τιμών που συνεχίζουν να υπάρχουν μεταξύ των γενετικά τροποποιημένων και των μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Βουλγαρία και Ρουμανία, μέσω αυτών περνάνε αυτές οι εισαγωγές. Και από την 1η Ιανουαρίου του 2014 θα ανοίξουν τα σύνορα και περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι θα μπορούν να κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη ελεύθερα και θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα προτιμούσα να είχε μπει 1,5 τόνος σόγιας στη θέση αυτών των ε, ε, ανθρώπων οι οποίοι θα έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κυκλοφορήσουν ελεύθερα. Γιατί βλέπετε ότι συνεχίζουμε και τα αυγά να τα παράγουμε με τον ίδιο τρόπο και να εισάγουμε γενετικά τροποποιημένη σόγια. Ευχαριστώ πολύ, Ρούμπιξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη. Έφτασα πολύ καθυστερημένος. Υπήρχε μια ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών και λυπούμε γιατί δεν μπόρεσα να ακούσω τον Υπουργό. Είμαστε γείτονες βέβαια, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και όσον αφορά την πραγματικότητα στη χώρα μου. Είμαι από τη Λετωνία. Έχω μεγάλη λοιπόν ελπίδα και εμπιστοσύνη στη χώρα σας. Ήδη από τη Σοβιετική εποχή η χώρα σας είχε μεγάλη ανάπτυξη στη γεωργία. Γνωρίζετε την διαχείριση του τομέα των αγροτικών θεμάτων. Έχετε μεγάλη εμπειρία και είμαι σίγουρος ότι θα προχωρήσουμε σε όλα τα εκκρεμή θέματα. Με τη δική σας Προεδρία. Εδώ και τρία χρόνια προετοιμάζουμε την μεταρρύθμιση της ΠΑΚ και Έχουμε πολύ συγκεκριμένα προγράμματα από το 2014 ως το 2020 η δική μου προσωπική άποψη συμβαδίζει με αυτή που παρουσίασαν οι εισηγητές. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν επεξεργαστεί τα θέματα αυτά, παρόλο που οι άμεσες πληρωμές φυσικά είναι χαμηλότερες από αυτές που ελπίζαμε και αυτό είναι κάτι που μας ε, στεναχωρεί. Η χώρα μου θα στηριχτεί στις προτάσεις σας και πιστεύουμε πραγματικά ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε και εμείς να εμπνευστούμε. Βεβαίως ε, δεν θα μπορέσετε να επεξεργαστείτε όλα τα θέματα και να ολοκληρώσετε όλες τις διαπραγματεύσεις και τις διαδικασίες μέχρι το τέλος της εξάμηνης προεδρίας σας, αλλά αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι το 7% της χρηματοδότησης δεν χρησιμοποιείται αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει καλύτερος έλεγχος, καλύτερη επιτήρηση της χρησιμοποίησης ε, των πόρων, των κονδυλίων, έτσι ώστε οι σπατάλες, αυτό το 7% να μην σπαταλάτε πλέον, αλλά να αρχίσει να χρησιμοποιείτε με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία για την ολοκλήρωση της Προεδρίας σας. Θα δώσω το λόγο στον Τζοβάνι Λαβία και κατόπιν στον Μισελ Νταντέν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς ε, και εγώ ε, θέλω να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία είπε η Προεδρία σχετικά με το πρόγραμμα του επόμενου εξαμήνου. Είμαι εισηγητής ε, της, ε, του οριζόντου κανισμού και γι' αυτό προφανώς ε, και θα υπογραμμίσω ότι είναι σημαντικό να σημειώσουμε πρόοδο. Σήμερα υπάρχει ε, πολιτική συμφωνία για το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Όσον αφορά τον οριζόντιο κανισμό και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουμε δύο θέματα. Το ένα θέμα αφορά την κρίση. Είναι προφανές ότι υπάρχουν προβλήματα γιατί η κρίση αυτή αφορά το κεφάλαιο 2, τη γραμμή 2 του προϋπολογισμού. Αυτό προϋποθέτει δημοσιονομική πειθαρχία και προϋποθέτει και σε άλλες περιπτώσεις την μείωση των άμεσων πληρωμών. Το θέμα λοιπόν όσο έχει κατατεθεί αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αναλυθεί, πρέπει να ε, εξεταστεί σε επίπεδο Συμβουλίου. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το θέμα, το Συμβούλιο και η Προεδρία, τι ακριβώς σκέπτονται από αυτού, πώς σκέπτονται να ελέγξουν το θέμα. Είναι σαφές ε, ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η θέση αυτή ήταν ε, πάντα επικριτική. Εμείς είχαμε και ένα απόθεμα για την ε, που είχαμε προβλέψει στον προπολογισμό, αυτό είχε χρηματοδοτηθεί ad hoc και όχι από τους ε, παραγωγούς. Ένα άλλο θέμα αφορά τη γεωργική ανάπτυξη. Είναι ένα θέμα που δεν το έχουμε εξετάσει μέχρι σήμερα. Το Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει κάποιες ε, τροπολογίες ε, με βάση αυτά ε, που επιθυμούν τα κράτη-μέλη, δηλαδή επιθυμούν υψηλότερες προκαταβολές, ενώ από την άλλη πλευρά εσείς στην αρχική σας εκτίμηση ε, σε επίπεδο Προεδρίας και σε ε, συμπεράσματα της 7ης και της 8ης ε, Φεβρουαρίου μειώσατε τους συντελεστές και τους φτάσατε σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο με στόχο προφανώς να μειώσετε τα εκταμιευόμενα κονδύλια. Είναι λοιπόν δύο τα ανοιχτά θέματα που πρέπει να εξετάσουμε και πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι η Προεδρία θα τοποθετηθεί από αυτόν. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο είναι εξίσου σημαντικό και νομίζω ότι από αυτού του θέματος ε, πρέπει ε, να υπάρξει ταχύτατα μια έρευνα, ένας έλεγχος. Πρόκειται για τα ε, μεταβατικά μέτρα. Γιατί κατ' ουσίαν ε, πρέπει να κλείσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, από αυτό το θέμα σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα έτσι ώστε από του χρόνου να γνωρίζουμε ακριβώς ε, τι θα ξεκινήσει σύντομα και τι θα αναβληθεί. Υπάρχουν θέματα σημαντικά όπως είναι η σύγκληση ανάμεσα στα κρατημέλη για τον πρώτο πυλώνα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι πως θα εξετάσουμε και τη μετάβαση ε, σε θέματα γεωργικής ανάπτυξης. Δεν ξέρω αν έχουμε πραγματικά τον απαραίτητο χρόνο τουλάχιστον με βάση τον νέο κανονισμό επί το οποίο έχουμε συμφωνήσει σε πολιτικό επίπεδο αλλά δεν έχουμε ακόμα το συγκεκριμένο κείμενο. Είναι λοιπόν σαφές ότι μας ενδιαφέρει ταχύτατα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, έχουμε από τις αρχές του 2014 μια κοινή γεωργική πολιτική για να μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία θα είναι νέα στοιχεία και τα οποία έκλεισαν υπό την Ιρλανδική Προεδρία. Πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, Τζοβάνι. Ο Μισελ ε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τον ε, Προεδρεύοντα και το πρόγραμμα εργασιών όπως το έχετε προκαθορίσει. Βεβαίως, ένα μεγάλο τμήμα της εργασίας σας θα είναι η ολοκλήρωση του πακέτου της κοινή αγροτικής ε, πολιτικής, της μεταρρύθμισης. Βεβαίως έχει επιτευχθεί η πολιτική συμφωνία. Το θέμα είναι βεβαίως ότι υπάρχουν ακόμα πολλές λεπτομέρειες οι οποίες είναι εκρεμείς. Στις 26 Ιουνίου το Κοινοβούλιο κατά κάποιο τρόπο βρέθηκε πρώτο τελεσμένου γεγονότος, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση του άρθρου 43.3 της συνθήκης. Με λίγα λόγια, οι Υπουργοί, το Συμβούλιο, αρνήθηκαν στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να εξετάσει κάποια ουσιαστικά εργαλεία για τη διαχείριση της κοινή αγροτικής πολιτικής, παραδείγματος χάρη διαχείριση κρίσης, και ιδιαίτερα την δυνατότητα παρέμβασης. Εγώ αυτό που είχα πει τότε είναι ότι το Κοινοβούλιο κοίταξε καταρχήν το συμφέρον όλων αυτών των γεωργών, των αγροτών, των φορέων, οι οποίοι θα έπρεπε να γνωρίζουν σχετικά νωρίς ποιο θα είναι το πλαίσιο στο οποίο καλούνται να δράσουν τα επόμενα χρόνια. Όμως το Συμβούλιο θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτές οι αποφάσεις και αυτή η διαπραγμάτευση είναι απογοητευτική για το Κοινοβούλιο και εκφράζομαι εδώ εξ ονόματος όλων των συναδέλφων και λέω ότι αυτή η ερμηνεία του 43.3, του άρθρου 43.3 της συνθήκης δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται επάπειρον στο μέλλον. Και εάν το Συμβούλιο επιμείνει σε αυτήν την ερμηνεία, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι θα έρθει μια στιγμή που θα εμποδίσουμε εμείς σαν κοινοβούλιο τις διαδικασίες. Πρέπει να συνεργαστούμε. Χρειαζόμαστε αμοιβαία εμπιστοσύνη και αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη σαφώς και χρειάζεται κοινή ερμηνεία της συνθήκης και μία συμμόρφωση και μία υπεύθυνη διαχείριση. Bene, grazie Michel. Continuiamo con eh, McGuinness. Πολύ ωραία, ευχαριστώ Μισελ. Κυρία Μαγκίνες, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που ήρθατε μας μιλήσατε. Πρώτα απ' όλα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, Τζοβάνι Λαβία πολύ σωστά είπε ότι έχει επιτεθεί η πολιτική συμφωνία σε την κοινωνική πολιτική. Αλλά τώρα θα πρέπει να δούμε στην πράξη πώ θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Η δε για σα, ε, κατά κάποιο τρόπο, ε, είναι πάρα πολύ σημαντική στο να εφαρμοστούν όλα αυτά και να περάσουν τα μηνύματα, να καταλάβουν περί τίνο πρόκειται η γεωργία μα. Νομίζω ότι ο Σεπτέμβριο θα είναι μήνα πάρα πολύ κρίσιμο. Άλλοι συνάδελφοι επίση έχουν ε, θεωρήσει ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική εδώ ε, πρόκληση για τα θέματα ε, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Οπότε θα πρέπει να δούμε ε, εμεί τι θέλουμε σε σχέση με την συναπόφαση και σε σχέση με τι αρμοδιότητε των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για να καλύψουμε το πολιτέ πλαίσιο, το δημοσιονομικό και τη γεωργία και φυσικά τους γεωργούς. Οπότε υπάρχει εδώ μια πάρα πολύ σημαντική πρόκληση, ούτως ώστε να μπορέσετε τα εν λόγω ζητήματα να τα προωθήσετε. Και φυσικά σας έχουμε σχετικά με αυτό καλή επιτυχία. Με ενδιαφέρει δε να μου πείτε, όσο και αν ακόμα είναι η αρχή της πορείας σας, πώς βλέπετε την εξέλιξη ε, αυτής της διαδρομής, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε την εκθεσιντές, ε, έχουμε την εκθεσιντές και θα πρέπει ε, τον έτρο δυνατό να λύσει κάποια ζητήματα. Άρα δεν θέλουμε να έρθει η λύση το Δεκέμβριο. Οπότε για πέστε μας πώς βλέπετε εσείς ε, ε, τα πράγματα, διότι κατά τη δική μου γνώμη αυτά όλα θα πρέπει να επιληθούν το Σεπτέμβριο. Και δεν είμαι βέβαιη ότι κάτι τέτοιο είναι ε, ρεαλιστικό. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς αν θα γίνει έτσι. Έχουμε επίσης σχετικές περικοπές και αν πρόκειται οι γεωργοί να ενισχυθούν λιγότερο από ε, την κοινότητα, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα γίνει με την αγορά, πώς θα έχουμε ε, υποστήριξη του εισοδήματός τους, για το πώς θα είναι δίκαιες οι ρυθμίσεις που αφορούν διατροφή και αλυσίδα. Και πάλι καλή επιτυχία. Πρόεδρος. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Η Ελίζαμπεθ και κατόπιν ο Αντιπρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε κύριε Υπουργέ ε, και θα ήθελα να σας ε, ευχηθώ μια επιτυχημένη Προεδρία. Βεβαίως άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά όλα αυτά που μας ε, είπατε σχετικά με τα θέματα που ενδιαφέρουν τη Λιθουανική Προεδρία. Για μένα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το τι θα κάνουμε κατά τους αμέσως επόμενους μήνες όσον αφορά ε, την κυνηγιορική πολιτική και την ε, κατανομή των ε, κονδυλίων. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που εκκρεμούν και για μας αυτό που μας απαγοήτευσε είναι ότι κατά τη διάρκεια της Ιλλανδικής Προεδρίας δεν ήταν δυνατόν να υπάρξουν συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις. Εμείς από πλευράς ε, Κοινοβουλίου θα επιμείνουμε στην εντολή που έχουμε λάβει και θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σας σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία εκκρεμούν ε, σε επίπεδο γεωργικής ανάπτυξης. Ε, όσον αφορά την κατανομή των κονδυλίων, αυτή είναι καθοριστική σημασία για μας. Το Κοινοβούλιο έχει δυνατότητε στο πλαίσιο της συναπόφασης και εν πάση περιπτώσει ε, εμείς θα υψώσουμε την φωνή μας όσον αφορά την διερευνητική εντολή. Και ως ε, προς τους ε, συντελεστές συγχρηματοδότησης αυτοί επηρεάζουν προφανώς τον, το σύνολο της Γεωργίας και θεωρώ ότι κυρίως ο εισηγητής έχει υποβάλει μια πάρα πολύ καλή πρόταση ε, που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας σας. Για μένα λοιπόν οι μεταβατικές διατάξεις είναι πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει ε, να προχωρήσουμε γρήγορα γιατί οι γεωργοί μας ε, χρειάζονται την ασφάλεια του προγραμματισμού. Κυρίως όσον αφορά την ενίσχυση των ε, επενδύσεων, οι γεωργοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια περιμένουν να στηριχθούν πλέον οι επενδύσεις γιατί αυτές οι επενδύσεις αφορούν σε μεγάλο βαθμό τις προδιαγραφές προστασίες που ισχύουν για τα ζώα. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε και θεωρώ ότι θα έχουμε μπροστά μας ένα πολύ ενδιαφέροντα Σεπτέμβρη. Πάντως σας εύχομαι καλή επιτυχία στην εφαρμογή των στόχων σας και οπωσδήποτε μια επιτυχημένη Λιθουανική Προεδρία. Ο κύριος Πόλσον και μετά ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ. Καλώς όρισε ο κύριος Υπουργό. Μικρή ή μεγάλη χώρα τελικά δεν έχει σημασία, διότι το θέμα είναι πώς κανείς προσεγγίζει τα θέματα. Τα ευρωπαϊκά, την Ευρώπη, την αναγκαιότητα να υπάρχει Ευρώπη. Τέλος πάντων θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μια Ευρωπαϊκή Προεδρία να μπορεί να φέρει σε αίσιο πέρα σε αυτή την μεταρρύθμιση. Γιατί ακόμη υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν, λεπτομέρειε που δεν είναι καθόλου εύκολες Οπότε τελικά ε, είναι θέμα συναπόφαση, είναι θέμα γεωργική πολιτική. Εγώ έχω αναλάβει έκθεση για την καλομεταχείριση των ζώων. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές επιτυχίες αυτής της δέσμης μέτρων που θα αφορούν την ε, διατροφική ασφάλεια. Άρα, υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές σε αυτό το ζήτημα και ίσως ε, το θέμα δεν είναι τόσο επίμαχο από πλευράς ε, πολιτικής. Όμως, από ε, τεχνικής αλλά και ε, πρακτικής υπάρχουν εδώ πολλές δυσκολίες και γι' αυτό και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον η Προεδρία έχει αρχίσει τις στο αναγκαίες επαφές. θα διανατούμε κατά πόσο να το μπορούμε τελικά να περιοριστούμε στα επιστημονικά στοιχεία και να επιλύσουμε και τις τυχόν πολιτικές προστριβές. Η Ευρώπη περνάει κρίση, βρίσκεται σε ύφεση, άρα θα πρέπει να εξελίξουμε την εσωτερική αγορά. τα ζωικά προϊόντα αλλά και τα ζώντα ζώα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχει ανοιχτό πνεύμα, ελευθερία, αλλά τι θα γίνει με τις επιζωτίες. Εδώ το ζήτημα είναι επίμαχο. Υπάρχουν διαφωνίες. Εάν θέλουμε να αποτρέψουμε τραγωδίες, όπως η αφρικανική νόσος και οι άλλες επιζωτίες που έχουν χτυπήσει θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε θα πρέπει να προλαμβάνουμε θα πρέπει οι γεωργοί κτηνοτρόφοι να έχουν την απαραίτητη γνώση ώστε να χτυπά το καμπανάκι του κινδύνου όσο γίνεται πιο νωρί. Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο οι γεωργοί εμπλίζουν τόσο επικίνδυνες καταστάσεις και που θα πρέπει να μπορούν να ανοιχνεύσουν την ευρωτυπησιότητα όταν χτυπήσει. Έχετε το λόγο πρόεδρε. Ε, συνάδελφε. Κοιτάξτε. Από όσα άκουσα χτες και όσα συζητήσαμε σήμερα, Ακόμα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Και εσείς επίσης, ως Προεδρία, κύριε Υπουργέ, από τι φαίνεται. Έχουμε προετοιμάσει κάποια πράγματα, αλλά θα πρέπει για να ολοκληρώσουμε τις προσπάθειές μας. Οπότε θα πρέπει ο κύριος Ντές να έρθει στη Λιθουανία να το πούμε εκεί. Και έτσι να λυθούν το πρόβλημα του κυρίου Ντέ. Ε, Τέλο, αυτό το λέω κάπω αστείο, μια που απευθυνθήκατε στον κύριο Ντέ προηγουμένω. Πάντω υπάρχει κάτι που δεν μα αναφέρεται στην αρχή, κύριε Υπουργέ. Κάτι για την ε, Γεωργία. Κάτι σε σχέση για τι ε, σχέσει μα επί του με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Διότι Έχουμε βέβαια κάποια άλλη επιτροπή που ασχολείται με τα θέματα εμπορίου, αλλά και τα εμπορικά ζητήματα είναι σημαντικά για μας, γιατί πολύ συχνά η Γεωργία είναι ο χαμένος τέτοιων ε, διαπραγματεύσεων. Είναι το θύμα των εμπορικών διαπραγματεύσεων όπως είπα. Ελπίζω ότι εσείς αυτή τη φορά θα έχετε μια διαφορετική, πιο κοινοτική προσέγγιση, πιο, θα έχετε πιο πολύ κατανόηση, στο Συμβούλιο. Θα είστε πιο φιλικός εισαγωγικά προς το Κοινοβούλιο και θα λάβετε υπόψη τις θέσεις μας. Άλλωστε αυτό το προβλέπει και η συνήθεια της Λισαβόνας. Καλή τύχη και πάλι. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πατρόν ναι, Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ μπορώ να συμφωνήσω με τους ε, συναδέλφους και εγώ σας ευχαριστώ. Είστε ευπρόσδεκτος και πραγματικά σας εύχομαι κάθε επιτυχία για το εξάμεινο της Προεδρίας της Λιθουανίας. Όπως ε, καταλάβατε, περιμένουμε πολλά από την Προεδρία της Λιθουανίας. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει, τα οποία είναι ακόμα μπλοκαρισμένα. Ελπίζουμε να φτάσουμε σε μια πραγματική αναθεώρηση της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής αυτό το εξάμεινο. Αναφερθήκανε οι συνάδελφοι σε κάποιες από αυτές τις υποθέσεις. Εμένα ιδιαίτερα με ενδιαφέρει ο τομέας του γάλακτος. Πρόκειται για το μεγαλύτερο θύμα αυτής της αναθεώρησης. Το Συμβούλιο δεν θέλησε να αλλάξει τίποτα στον τομέα αυτό. Σε σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα στην κοινή οργάνωση των αγορών. Υπάρχει το πακέτο για το γάλα και υπάρχει βεβαίως και το μέλλον του τομέα. Αν κοιτάξουμε το παρελθόν, διαπιστώνουμε ότι το μέλλον δεν είναι λαμπρό για τον τομέα αυτό. Δεν υπάρχουν καν προτάσεις οι οποίες να μας δίνουν κάποια ελπίδα. Υπάρχει η έκθεση για την παραγωγή του γάλακτος, υπάρχουν κάποιες προτάσεις πολύ συγκεκριμένες για τις πολύ απομακρυσμένες περιοχές, για τις ορεινές περιοχές, αλλά Πρόκειται για μια παραγωγή που είναι καθοριστική σε κάποιες περιοχές και πραγματικά επαναλαμβάνω ότι το θέμα αυτό ξεχάστηκε, θυσιάστηκε θα έλεγα στην αναθεώρηση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ποιες είναι λοιπόν οι προθέσεις σας, ποιες είναι οι προθέσεις της Λιθωνικής Προεδρίας. Πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος γνωρίζει κρίσεις κυκλικές κατά κάποιο τρόπο. Τι θέλετε λοιπόν να κάνετε και τι προτίθεστε να κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον ε, Υπουργό, ο οποίος θα απαντήσει. Έχουμε χρόνο, μπορείς να απαντήσεις σε όλες τις προτάσεις ε, των συναδέλφων. Υπάρχουν πολλές προσδοκίες τις οποίες έχει το δικό μας το Κοινοβούλιο σε σχέση ε, με την ολοκλήρωση αυτή την τόσο σημαντική διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική για μας ε, και για λόγους αρχής. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποκλειστεί από την διαπραγμάτευση των τελευταίων στοιχείων της ε, μεταρρύθμισης ε, δεν μπορεί να αποκλειστεί το Κοινοβούλιο επειδή το Συμβούλιο μπλοκάρισε κατά κάποιον τρόπο την απόφαση των Υπουργών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα ε, μας προσφέρονται όλες οι δυνατότητες για να προχωρήσουμε, να συμμετέχουμε και ελπίζουμε να κλείσει το θέμα κάτω από τη δική σου την Προεδρία. Ελπίζω, λοιπόν, ε, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μεταρρυθμίσεων γιατί η Ευρώπη περιμένει όλα αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα. Θέλουμε να ενημερώσουμε τους ε, γεωργούς μας και να αρθούμε στο ύψος των ε, περιστάσεων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βιτζίλιους, και έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, για την επιθυμία της Προεδρίας. Σημείωσα όλα όσα είπατε, τα σχόλιά σας και φυσικά και θα τα λάβουμε υπόψη. Θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η επιτυχία των αποφάσεών μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αμοιβαία συνεννόηση και κατανόηση, από την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Χρειαζόμαστε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης και είναι αυτό στο οποίο πραγματικά προσβλέπουμε για τους επόμενους έξι μήνες. Αμοιβαία εμπιστοσύνη, ένα κλίμα συνεργασίας το οποίο θα μας οδηγήσει σε καλά κοινά αποτελέσματα για τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε σήμερα σωστή βάση θεμέλια στο μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής. Αυτό μπορούμε να το οικοδομήσουμε από κοινού. Και θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Μας πιέζει ο χρόνος βέβαια, γι' αυτό και θα επικεντρωθώ στα κύρια σημεία που επανέλαβαν πολλοί ομιλητές. Σίγουρα θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε στο μέλλον σε πιο άτυπες συναντήσεις. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να εστιάσω στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πολύ πρόσφατα πετύχαμε μια συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ολοκληρώθηκαν και ήρθε η ώρα να λύσουμε επιμέρους θέματα που αφορούν τις προοπτικές του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου και σας υπόσχομαι ότι για όλα τα άλλη τα εκρεμή θέματα θα συνεργαστούμε γνωρίζω ποια είναι η εντολή σας και εσείς γνωρίζετε ποια είναι η δική μου εντολή από μέρους του Συμβουλίου. Γνωρίζετε επίσης τις πρόσφατες προτάσεις στον τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων. Δεν έχω απολύτως καμία νέα εντολή. Πρέπει λοιπόν να δούμε πως οι κοινέ μας αποφάσεις θα εξελιχθούν επικοδομητικά. Αυτό μπορώ να το κάνω. Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης της κοινή αγροτικής πολιτικής εμπεριέχει πολύ τεχνική εργασία. Η ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου επίσης εμπεριέχει τεχνικά τμήματα. Θα γίνουν συναντήσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων για το χτένισμα των κειμένων και πιστεύω πραγματικά ότι μέσω αυτών των επικοδομητικών συζητήσεων θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τα επιμέρους ζητήματα που παραμένουν εκρεμή και να δώσουμε εγγυήσεις για το μέλλον. Και τώρα θα θέλω να μιλήσω για την μεταβατική περίοδο, για τον κανονισμό που είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο οποίος θα πρέπει να υιοθετηθεί στο άμεσο μέλλον. Ο κύριος Ντές είπε πολύ σωστά ότι και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ότι έχουμε την ευθύνη να υλοποιήσουμε αυτή την υποχρέωσή μας έτσι ώστε οι αγρότες στην Ευρώπη να μην βρεθούν σε ένα κενό το 2014. Και για την κτηνοτροφία και για τη γεωργία η μεταβατική αυτή περίοδος είναι εξαιρετικά σημαντική όσον αφορά την υγεία, την ευημερία των ζώων, όσον αφορά την παραγωγή των, ε, στα ορνηθοτροφία, οι οτόκες όρνηθες, οι ρυθμίσεις δεν είναι αν θέλετε, οι ιδανικές. Το πρόβλημα είναι όμως ότι αυτά που έχουν αποφασιστεί δεν εφαρμόζονται. Η Προεδρία της Λιθουανίας θα προσπαθήσει λοιπόν να υλοποιήσει αυτές τις αποφάσεις, κάτι το οποίο θα πρέπει να ισχύσει σε όλη την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τη σόγια και τους τροποποιημένους γενετικά οργανισμούς. η γενετικά τροποποιημένη σόγια είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζουμε. Χρησιμοποιείται για ζωοτροφές, όχι μόνο για τα πτηνά, όχι μόνο για τις όρνηθες, αλλά και για πολλά άλλα ζώα. Η διατροφική αλυσίδα λοιπόν θα πρέπει να ελέγχεται έτσι ώστε να υπάρχει σωστή ενημέρωση για τους καταναλωτές. Όσον αφορά τη δική μου χώρα, η έλεγχη είναι εξαιρετικά αυστηρή όσον αφορά τη χρήση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και ξέρω ότι και άλλα κράτη-μέλη το κάνουν. Η ευθύνη είναι δική μας, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, πρέπει να υπάρχει ταχύτατη ανταλλαγή πληροφοριών για τα θέματα αυτά. Και βεβαίως θα πρέπει να βρούμε και άλλες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά τις ζωοτροφές και όσον αφορά την αντικατάσταση της γενετικά τροποποιημένης σόγιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι θέμα επιστημονικό, υπάρχουν ε, επιστημονικές αναλλακτικές προτάσεις και σίγουρα θα πρέπει να στηρίξουμε προγράμματα τα οποία να προωθήσουν αυτές τις εναλλακτικές λύσεις. Και βεβαίως οι προβλέψεις αυτές εμπεριέχονται στον προϋπολογισμό Κάνω εδώ μια έκκληση για δημοσιονομική πειθαρχία. Το αποθεματικό του προϋπολογισμού περιέχει κάποιες δυνατότητες και στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου υπάρχει δυνατότητα πολύ περιορισμένη. Οι αρμοδιότητές μας επίσης είναι πολύ συγκεκριμένες και εδώ θα πρέπει να εναρμονιστούμε στις διατάξεις της Λισαβόνας. Η αποστολή μας είναι να βρεθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό νομίζω θα γίνει μετά την πρώτη ανάγνωση Επιτρέψτε μου επίσης να αναφέρω τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες συνεχίζονται για το πακέτο της αναθεωρήσης της ΚΑΠ. Καταφέραμε να υιοθετήσουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Όσον αφορά πάντα τις διατάξεις ε, της ε, Λισαβόνας. Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω όσον αφορά τον κανονισμό για την υγεία των ζώων, την ευημερία των ζώων, μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας της χώρας μου. Όσον αφορά τις νόσους, τις επιζωτίες, Ο κατάλογος αυτών των ε, νόσων είναι κάτι που θα γίνει από τις ε, ομάδες των ε, εμπειρογνωμόνων, οι οποίες σε τεχνικό επίπεδο έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία του θέματος και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την κίνημα συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά το ίδιο αυτό θέμα, την ευημερία των ζώων, επιτρέψτε μου να σας πω ότι στην χώρα μου στη Λιθουανία δίνουμε μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό και και πιστεύω ότι αυτή η σημασία θα πρέπει να είναι κοινή σε όλες τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνω μια έκκληση προς όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να φτάσουμε σε κοινό επίπεδο για την ευημερία των ζώων, βασιζόμενη σε επιστημονικά δεδομένα. 28 και 29 Σεπτεμβρίου οργανώνουμε στη Λιθουανία μία συνάντηση για την ευημερία των ζώων, για τις ζωοτροφές και θα είμαι παρόν σε αυτήν την συνάντηση. Σας προσκαλώ λοιπόν όλους στην συνάντηση αυτή. Δύο λόγια τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώτος γύρος, το πρώτο επίπεδο των διαπραγματεύσεων ξεκίνησε στη Ουάσιγκτον. Η σημασία αυτών των διαπραγματεύσεων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερεκτιμηθεί. Ελπίζω να εξελιχθούν όλα ομαλά. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και φυσικά εμείς θα επιμείνουμε για πολύ αυστηρά πρότυπα όσον αφορά τα φυτά, όσον αφορά την υγεία των ζώων. Σκοπός μας είναι όμως ταυτόχρονα να υπάρξει εξάλληψη των ε, εμπορικών εμποδίων. Έρχομαι τώρα στο γάλα. Το πακέτο αυτό έχει ολοκληρωθεί με την συμφωνία και την κοινή οργάνωση της αγοράς στις 24 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες σε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου θα συζητηθεί το θέμα αυτό και πιστεύω ότι εκεί θα μπορέσουν να βρεθούν οι λύσεις που είναι απαραίτητες για να καλυφθούν οι αδυναμίες του τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ ε, επικοδομητικά σας σχόλια, για τις ερωτήσεις σας, για τη φιλοξενία σας και ελπίζω ότι τους επόμενους μήλες θα συνεχίσουμε την επικοδομητική μας συνεργασία. Πολύ ωραία και εμείς ε, Ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον Δετζίλιο Σεγιούκνερ. Ε, πράγματι θα έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά και ειλικρινά ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσουμε ε, υπό τη δική σας προεδρία όλα αυτά τα σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να διαπραγματευτούμε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την μεταρρύθμιση της ΠΑΚ. Συνάδελφοι, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή στην ε, ακρόαση για το μέλλον των των απορροκυπευτικών στην Ευρώπη, θέλω να σας πω μερικά πράγματα για να σε ενημερώσω. Καταρχήν το ότι ο γενικό μα γραμματέας, ο κύριος Γκέρλ Κάλπ, μας αφήνει και αυτή είναι η τελευταία Επιτροπή γεωργία στην οποία είναι παρόν, γιατί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου και πριν από αυτήν θα, πάει, θα βγει στη σύνταξη όπως ξέρετε ίσως μερικοί από εσά. Θέλω λοιπόν εξ όλων να τον ευχαριστήσω κυρίως για τα δύο τελευταία χρόνια που περάσαμε μαζί ε, και είδαμε ότι τα χρόνια αυτά μπορέσαμε να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Ε, είχε πάντα υπομονή ε, και επέδειξε ιδιαίτερη προσοχή σε όλους τους εισηγητές. Νομίζω λοιπόν ότι κατορθώσαμε πολύ καλά αυτή τη μετάβαση προς την συναπόφαση και προς την ανάλυση περισσότερων ευθυνών και αρμοδιοτήτων ως Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω το χρωστάμε ε, συγχαρητήρια και του ευχόμαστε καλή τύχη, κάθε καλό ε, σε μια καινούργια περίοδο που δεν θα έχει πια τόσες ευθύνε ε, όσο είχε, όσους είχε τον τελευταίο καιρό. Και με πάση περιπτώσει θα έχει την ευκαιρία να χαρεί την οικογένειά του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα λοιπόν... Ο κύριος Ντες ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους του ΕΛΚ ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ θερμά τον Γκέρχαρτ Κάλκ. Η συνεργασία μαζί του, η μακροχρόνια συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή. Ε, κοιτάξτε, σου έχω φέρει και ένα δωράκι με την αφιέρωση. Αξιότιμη κύριε Κάλπ, ονόματός μου και εξ ονόματος του ΕΛΚΑ της Επιτροπής Γεωργίας σε ευχαριστούμε για την πολύ καλή συνεργασία, την αγαστή συνεργασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Θαύμαζα πάντα ε, την υπομονή σας, την ηρεμία σας, την υφαλιότητα σε αυτή την καινούρια φάση της ζωής σας, υγεία, ευτυχία και ε, μια υποσημείωση. Ε, σου εύχομαι με το βιβλιαράκι αυτό να ευχαριστηθεί σε αυτά που γράφει ο φίλος μου ο Τσέπφλ από τη Βαβαρία. Και επιτρέψτε μου κύριε Κέτλ να σας δώσω αυτό το δωράκι, το βιβλίο. Ε, πολύ ωραία. Ο Λουίς Κάπουλα Σάντος ε, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κι εγώ να πω δύο λόγια για να αποχαιρετήσω τον ε, γραμματέα μας, ο οποίος είναι μαζί μας εδώ και 10 χρόνια, εξ ονόματός μου και εξ ονόματος όλων των συναδέλφων τον ευχαριστώ για την εργασία του, για την αφοσίωσή του, γιατί με αυτόν τον τρόπο μας δείχνει πώς μπορεί ένας υπάλληλος να είναι διακριτικός και αποτελεσματικός. Γενικό ε, ε, Γραμματέα, εκείνο Πάτρικ Πατσόλα. Βεβαίω θα πρέπει να περιμένουμε τον επίσημο διορισμό του νέου ε, Γενικού Γραμματέα. Δίνω όμω το λόγο στον Τζορτζ που τον ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ από πλευράς Εργατικού Κόμματος και εγώ να σας ευχαριστήσω για όλα όσα μας είπατε και που μας ανεχτήκατε. Γιατί ιδίω την τελευταία διετία η μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική ήταν ε, ένα, ένα άθλος άθλο. Ε, και σας ευχαριστούμε που μας βοηθήσατε σε όλη αυτή την διαδρομή της συναπόφασης και προσδώσατε αξιοπιστία σε όλη την ευρωτευτική ομάδα. Και πάλι ευχαριστώ που κρατήσατε έτσι στιβαρά το τιμόνι αυτή τη διαδικασία. Τζόσεφ, ευχαριστώ. Θέλει και ο Μάρτιν να... ή ο Τζιμ να πει δύο λόγια. Μάρτιν. Με μεγάλη χαρά εργαστήκαμε μαζί σου τα τελευταία χρόνια αυτές οι 7.000 τροπολογίες που υποβάλαμε με τι ηρεμία και αποτελεσματικότητα τις αντιμετώπισης και πραγματικά ήσουν δεξιοτέχνης στη διαχείριση αυτών των θεμάτων. Μπράβο. Όσον αφορά την αναθεώρηση, ναι, ας είπες πρέπει να ξεκινήσουμε από νωρίς και κατόπιν να ξεκουραστούμε στα πουνά σου. Εύχομαι κάθε καλό και ελπίζω που και που να έρχεσαι εδώ στις Βρυξέλλες να μην μας ξεχάσεις τελείως. Ελπίζω ότι μπορούμε που και που να βασιζόμαστε στην παρουσία σου, στην στήριξή σου και σου εύχομαι κάθε καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριο Jim. Πρόεδρε, είναι απόφραση μέρα αυτή. Τέλο πάντων, όπως και όλοι οι άλλοι, και εγώ να ευχηθώ ε, καλή συνέχεια ε, και καλή σύνταξη τέλο πάντων, αλλά δεν νομίζω ότι ε, δείχνει ότι είσαστε για σύνταξη τόσο κάνατε για προσπάθειά σας για την ΚΑΠ και τη μεταρρύθμιση. Ήταν μεγάλη αυτή η πορεία που κάναμε μαζί. Και Μαρία βλέπω, είναι εδώ που και εκείνη μας συνόδευσε σε αυτή τη ε, διαδρομή. Θυμάστε και εκείνη την αποστολή που κάναμε στη Βραζιλία για το βόλιο κρέας. Ε, η Λουίζ επίσης μας συνόδευσε. Και περάσαμε πολλά, πολλά και δύσκολα με τους ε, αγρότες, με τους πολιτικούς. Πολύ πολύ σκληρή ήταν η μάχη που δώσαμε στη Βραζιλία. Δεν ήταν σαν κυριακάτικη εκδρομή όπως πολλές φορές νομίζουν ότι κάνουμε στις αποστολές ξενύχτια, εργασίας, συνεδριάσεις ατελείωτες, αλλά στο τέλος Πήγαμε σε εκείνο το υπερμοντέρνο σφαγείο. Μας κεράσαν. Μοσχαρίσιο. Ε, και θα να, να πάρουμε και μαζί μας λίγο. Ε, τέλος πάντων, οι αναμνήσεις είναι εξαιρετικές από τη συνεργασία μας και από εσά και από όλο το επιτελείο σας και νομίζω, Πρόεδρε, ότι θα έχουμε και τις ε, στο μέλλον όλοι. Ωραία. Συνάδελφοι, ένα λεπτάκι, θα κάνουμε διάλειμμα, θα αποχαιρετήσουμε τον Βυργίλιο και ευθύσαμε αμέσως μετά αρχίζει για το προκυπευτικά η ακρόαση. Λοιπόν, συνάδελφοι, φτάσαμε στο τελευταίο σημείο στην ε, ακρόαση σχετικά με τα απορροκυπευτικά στην Ευρώπη, στρατηγική για την ανάπτυξη. Και τώρα έχουμε ε, ακρόαση για το μέλλον ε, αυτού του τομέα στην Ευρώπη, η στρατηγική ανάπτυξη. Σε όλη αυτή την ακρόαση την έχει οργανώσει η κυρία Μέκιντάιν και όπως ξέρετε ε, η κυρία Μέκινταν είναι η συγγήτριά μας. Πρέπει λοιπόν να καταθέσουμε προτάσεις σε σχέση με αυτή την τόσο σημαντική ακρόση. Ο τομέας των απορροκυπευτικών, όπως γνωρίζετε ε, περιλαμβάνει ε, τα βρόσιμα εκτός από τα διακοσμητικά φυτά και ένα σημαντικό κομμάτι της γεωργίας. Υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις σε επίπεδο κλιματικής αλλαγής και πρέπει όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε όπως και άλλα εμπόδια. Όλα αυτά είναι ε, σημαντικά θέματα για τον τομέα και για την γεωργία. Έχω λοιπόν τη μεγάλη χαρά εδώ να μπορώ να φιλοξενήσω τέσσερις ε, διακεκριμένους ε, ομιλητές, Έντονι Σνέλ, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος ε, της Εθνικής Ένωσης Γεωργών του Ηνωμένου Βασιλείου και ασχολείται ειδικά με τα οποροκυπευτικά, ο κύριος George Μπρότονς, ο οποίος είναι πρόεδρος ε, της ε, Ομοσπονδίας των Ισπανών, πάλι για τον ίδιο τομέα, τον κύριο Ντονάτο Λαμπάτε, που είναι μέλος του Συμβουλίου του ΣΟΠ, που είναι η Ένωση Οποροκυπευτικών και τέλος, ο κύριος Δίκφριτ Σόλτς, ο οποίος είναι ε, γενικός γραμματέας ε, ε, της, των αποκερπευτικών μια συγκεκριμένη ένωση αποκερπευτικών στη Γερμανία. Και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους σας. Όλοι έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας και πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συνάδελφό μας την Αντέα. Παρακαλώ Αντέα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Λέει η Άννη Μακιντάερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά. Έχουμε σήμερα αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για το πολυκυπευτικά. Οπότε και θα μπορέσουμε να ακούσουμε κάποιους πραγματικά ειδικού ή στο θέμα. Τα προκυπευτικά είναι ιδιαίτερα περίπλοκος τομέας. Και μάλιστα ε, δεν τον καταλαβαίνω τόσο καλά, αλλά τώρα που Μα απασχολεί όλο ένα και περισσότερο η διατροφική ασφάλεια. Ο κλάδο των προεκπαιδευτικών έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Και ε, ας πούμε από το δικό μου χωριό εκεί στο West Midlands, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, ενδεικτικά ε, είναι κάτι το οποίο δείχνει, το ενδιαφέρον δηλαδή εκεί του, του, τόπου μου, πόσο σημαντικά είναι τα προεκπαιδευτικά. Πολλές οι προκλήσεις, πολλές και οι ευκαιρίες που προσφέρονται. Και είμαστε ο αθλητή παγκοσμίω. Αλλά είμαστε και ο αθλητή εκτός από την παραγωγή και στις εισαγωγέ. Οπότε ε, θα πρέπει να δούμε το ότι έχουμε κάμψει στην ε, προσφορά και επομένως ε, θα πρέπει να υπάρξει κάποια ανάπτυξη στον κλάδο. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Ανάπτυξη και έρευνα μπορεί να βοηθήσουν πόροι, παραγωγικότητα και υπάρχουν και άλλα ζητήματα των καλλιεργητών, θέματα ενεργειακού κόστους, προστασίας της παραγωγής, ε, ίδρευση, κατάρτιση, ε, προστασία του περιβάλλοντος, γιατί πρέπει να παραγάγουμε περισσότερα από λιγότερα. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και θα πρέπει όλα αυτά να τα καλύψουμε την έκθεσή μας. Πάντως, είναι πάρα πολύ θετικό το ότι θα ασχοληθεί η Λιθουανική Προεδρία το φθινόπωρο. Και επίσης η έκθεσή μας θα βοηθήσει. Αλλά και η σημερινή μας ακρόαση πρόκειται επίσης να ενημερώσει. Bardzo dziękuję pani poseł sprawozdawcy. Przechodzimy w tej chwili do wysłuchania. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Συγγήτρια. Προχωρούμε τώρα στην ακρόαση. Κύριος Αντώνη Σνέλ θα λάβει τώρα το λόγο. Good morning everybody. Uh, my name's Anthony Snell. I'm, I'm... Καλημέρα. Λέγομαι Άντωνη Σνέλ και είμαι αντιπρόεδρος της ε, Ένωσης Οπροκυπευτικών NFU Θα ήθελα να σας μιλήσω για την περιοχή των West Midlands, των δικών Midlands, στο Hertfordshire, από όπου προέρχομαι. Πρόκειται για μια περιοχή με μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Η Άνθια είναι μεγάλος υποστηριχτής ε, της παραγωγής οποροκυπευτικών και περίπου 2.000 τόνοι 6.000 τόνοι βατόμουρων, ε, φράουλες ε, και μούρα παράγονται στην περιοχή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να ελέγξουμε όλη την διατροφική αλυσίδα και να εφοδιάσουμε την αλυσίδα αυτή με σοβαρούς ε, ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καταρχήν και σε αυτή τη φωτογραφία βλέπετε παιδιά από σχολεία που επισκέπτονται τα αγροκτήματά μας με σκοπό να πλησιάσει ο καταναλωτής την παραγωγή. Χρειαζόμαστε μια ευέλικτη και ε, εποχιακή δυνατότητα πρόσληψης ε, εργαζομένων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ξαναδούμε αυτό το ε, ισχύον σύστημα για την εποχιακή εργασία, ιδιαίτερα για τα αγροκτήματα. Στην περιοχή μας λοιπόν παράγουμε 30% της παραγωγής πατάτας, 40% των φρούτων, των μήλων, 60% και 35% των βατόμουρων της ε, χώρας μας. Πρόκειται για μια σημαντική λοιπόν ε, ε, περιοχή που παράγει 50% περίπου της συνολικής παραγωγής. Είναι μια μικρή περιοχή και 650.000 ε, ευρώ είναι η προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς. Είναι ένας μεγάλος λοιπόν σημαντικός τομέας, επίσης και για τον τομέα του γάλατος και των δημητριακών. Θεωρώ ότι ο δικός μας τομέας, το τομέας των ε, κυπευτικών είναι εξαιρετικά σημαντικός, αλλά δεν εστιάζεται η προσοχή αρκετά σε αυτόν. Πέρσι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, ε, ένα δύσκολο έτος για τους παραγωγούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, για όλους τους τομείς των ε, οποροκυπευτικών, με μειωμένα κέρδη, μειωμένη παραγωγή, που βεβαίως οφείλεται τις καιρικέ συνθήκες, με μείωση των πωλήσεων, με μείωση των κερδών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε τις περισσότερες βροχές τα τελευταία 100 χρόνια με πολύ καθυστερημένη άνοιξη και το 2012 αυτό το πλεόνασμα βροχής, βροχοπτώσεων, κάτι που οδήγησε σε σημαντική η επιδείνωση της ποιότητας και θεωρούμε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα χρειαστούμε τουλάχιστον 20% παραπάνω αποθηκευτικούς χώρους για τα πλεονάσματα μέχρι το 2020. Ο απρόβλεπτος καιρός είναι κάτι που σίγουρα θα αποτελέσει πρόκληση για το μέλλον. Παρόλα βεβαίω όλα αυτά, είμαστε πολύ αισιόδοξοι στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον τομέα αυτό. Προς το παρόν ο καιρός είναι πολύ καλός και στον τομέα μας βλέπουμε η παραγωγή να αυξάνεται, τα κέρδη να αυξάνονται και όλα τα τμήματα της αλυσίδας, της εφοδιαστικής αλυσίδας να εμπλουτίζονται. Είμαστε ένας τομέας ο οποίος βεβαίως θα πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του και θα πρέπει ο τελικός καταναλωτής να πλησιάσει τον παραγωγό. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες του ΕΒ. Η υγιεινή διατροφή και η αύξηση της κατανάλωσης σε λαχανικά και φρούτα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή, κάτι το οποίο είναι καλό για την υγεία. Υπάρχει σημαντικό κέρδος για όλους. Και δεν θα αναφερθώ μόνο στο οικονομικό κέρδος. Όσον αφορά την αύξηση της παραγωγής και την αύξηση των κερδών, αυτό βεβαίως είναι κάτι που θα πρέπει να ακολουθήσει πολλά στάδια. Εδώ βλέπετε τη νέα σήμανση της βρετανικής ντομάτας. Το ίδιο έγινε και για τα φασολάκια και για τα μανιτάρια το 2012. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εξέβρεσης εδάφους στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον οποίο να μην είναι μολυσμένο από λιπάσματα για τη βιολογική καλλιέργεια. Στην ε, έκθεση που δημοσιεύσαμε το 2012 παρουσιάζουμε όλα αυτά τα στοιχεία, κάτι που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών. Παραγωγών σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας. Υπάρχει σήμερα μια έντονη συζήτηση όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της αλυσίδας. Περισσότερη διαφάνεια, πιο αυστηρή έλεγχη. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε την κατανομή της τιμής για το 2011 και βλέπετε το κομμάτι που, του κέρδους, της τιμής που πάει κατευθείαν στο λιανικό εμπόριο με κόκκινο χρώμα. Και βλέπετε ότι η απειλή στην Ευρώπη είναι να μειωθεί το μερίδιο των οποροκυπευτικών που παράγονται στην Ευρώπη στα πολυκαταστήματα, στα σούπερ μάρκετ και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε δυστυχώς να αυξάνεται σαν τάση. Ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι οι ενώσεις των παραγωγών να ξεκινήσουν μια νέα εκστρατεία ενημέρωσης με συγκεκριμένες πληροφορίες για τον καταναλωτή όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων και τον τρόπο παραγωγής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν ξεκινήσει οι διαβολεύσεις όσον αφορά την στρέβλωση του ανταγωνισμού και μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία για μια αξιολόγηση των πρακτικών που εφαρμόζονται και ισχύουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό είναι κάτι που βεβαίω θα πρέπει να ξεπεράσει το Ηνωμένο Βασίλειο και να επεκταθεί σε όλες τις χώρες. Είμαι μέλος ενός συνεταιρισμού Berry Gardens παράγουμε φρούτα για όλη μας την περιοχή. Η προστιθέμενη αξία αυτών των, ε, αυτής της παραγωγής είναι κάτι το οποίο έχει αυξηθεί προς όφελος βεβαίως και του καταναλωτή αλλά και των παραγωγών. Θεωρούμε πραγματικά ότι σήμερα μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της παραγωγής μας παρόλο που θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε ακόμα πολύ προσεκτικοί και στον Ηνωμένο αλλά και σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά την ε, αύξηση της παραγωγικότητας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φτάσουμε σε επίπεδα παραγωγής που να μπορούν να απορροφηθούν από την αγορά. Χρειαζόμαστε καινοτομία, χρειαζόμαστε έρευνα, νέες τεχνικές για την αποθήκευση, για τη μεταφορά, κάτι το οποίο σήμερα δεν στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπουμε σήμερα ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μείωση των παραγωγών και όσον αφορά τους συνεταιρισμούς και τις ενώσεις παραγωγών θα πρέπει να αλλάξει η τάση και να αντιστραφεί ο σημερινός προσανατολισμός. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι Βρετανοί παραγωγοί να μπορούν να συμμετάσχουν σε εταιρικέ σχέσεις με άλλους παραγωγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό βεβαίως και σε άλλους τομείς της παραγωγής, όχι μόνο στα οποροκυπευτικά, στα φρούτα, αλλά και στον τομέα του γάλατος, κάτι το οποίο είναι σήμερα απαραίτητο. Ανησυχούμε γιατί βλέπουμε κάποιες τροπολογίες ε, την ε, πρόταση για τα όπορο κυπευτικά που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποσυρθούν ή να αλλάξουν. Θεωρούμε ότι οι οργανώσεις των παραγωγών θα πρέπει εδώ να εισακουστούν. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην προστασία της καλλιέργειας. Όσον αφορά καταρχήν τις ε, μέλισσες, ξέρετε ότι για τους παραγωγούς οι μέλισσες είναι απαραίτητες. Αγαπάμε και θέλουμε να προστατεύσουμε τις μέλισσες, κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η πρόσφατη απόφαση της ε, Επιτροπής να απαγορευτούν για δύο χρόνια οι ουσίες που χρησιμοποιούνται και οι οποίες έχουν αρνητικές συνέπειες στις μέλισσες δείχνει πόσο λανθασμένη κατεύθυνση είχε λάβει η αγροτική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει σήμερα να μην βασιζόμαστε σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά στην κοινή γνώμη και στην ιδεολογία. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τον κανονισμό για τα φυτοφάρμακα και τα ζυζανιοκτώνα, έτσι ώστε να μην βρεθούμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στα επόμενα χρόνια. Η ασφάλεια της παραγωγής τροφίμων είναι καθοριστική και σε καμία περίπτωση οι Ευρωπαίοι παραγωγοί δεν θα πρέπει να βρεθούν σε μια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τον ανταγωνισμό από τις τρίτες χώρες. Θέλω λοιπόν να είμαι θετικός, θέλω να είμαι αισιόδοξο, αλλά ένας παραγωγός θα πρέπει σήμερα να μπορεί να βρίσκεται σε μια οικονομία ανταγωνιστική, σε ανάπτυξη λύσεων και στρατηγικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο η παραγωγή θα πρέπει να μπορεί να παράγουν, να είναι ανταγωνιστική και να ζουν από την εργασία τους με σκοπό να παράγουν ασφαλή τρόφιμα στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες όπως αυτή η σημαντική έκθεση και οι σημαντικές οργανώσεις της ε, γεωργικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα αιτήματα του οποροκυπευτικού τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα τώρα να προσθέσουμε το ότι ο κ. Νέλ είναι αντιπρόεδρος του Εθνικού Φορέα Γεωργών στη χώρα του. Και πάλι ευχαριστούμε κ. Σνέλ. Θέλω να δώσουμε τώρα τον λόγο στον ε, Ισπανό εκπρόσωπο των παραγωγών και εξαγωγών οπωροκυπευτικών, τον Χόρχε Μπροτόνς. Buenos días. Señor presidente del Comité de Agricultura y de... Καλημέρα σας. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπέθρου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι της Βουλή Επιτροπής και εκπρόσωποι του κλάδου των προκυπευτικών. Τα προκυπευτικά στην Ισπανία και σε πολλές ε, περιοχές είναι ο πυρήνας της ε, γεωργικής οικονομίας διότι εκπροσωπούν την ε, πλειοψηφία, το μεγαλύτερο ποσοστό της ε, παραγωγικής δραστηριότητας και αυτό αφορά και τα οικονομικά μεγέθη αλλά και από πλευράς απασχόλησης. Επίση, βοηθούν πάρα πολύ όσον αφορά την διατροφική ασφάλεια και μια υγιεινή διατροφή. Στην Ισπανία μιλάμε για το 55% τη γεωργική παραγωγή και αυτό επικεντρώνεται σε κάποιε περιοχέ όπου έχουμε ανεργία η οποία είναι πάνω από 30% και εκεί όπου έχουμε ανεργία των νέων πάνω από 50%. Επομένω, η κοινωνική λειτουργία του κλάδου αυτού είναι πάρα πολύ βασική διότι εκπροσωπεί το 50% τη απασχόληση στον τομέα τη γεωργίας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία νομίζω ότι δεν έχει ληφθεί ε, ακριβώς ε, υπόψη όπως έπρεπε όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική. Οπότε για τώρα συνεχίζουμε κάποιες πολιτικές οι οποίες μέσα σε μια συγκυρία κρίσης όπως σήμερα δεν επικεντρώνουν τις προσπάθειες αλλά και τις ενισχύσεις εις την παραγωγική δραστηριότητα αλλά και εις την απασχόληση στον γεωργικό τομέα. Και σαν συνέπεια τούτου ο κλάδος ε, αντιμετωπίζει τώρα προβλήματα τα οποία θα μπορούσα να τα εστιάσω σε τρία τεινά. Πρώτα πρώτα εμπορική πολιτική, δεύτερον γεωργική πολιτική και τρίτον έρευνα. Στην εμπορική πολιτική έχουμε μια παγκοσμιοποίηση η οποία είναι ασυμμετρική ή ασύμμετρη όσον αφορά τι αγορέ. Έχουμε την ε, ολοκληρωτική, ε, το ολοκληρωτικό άνοιγμα τη κοινοτική αγορά όσον αφορά τι εισαγωγέ. Οπότε τώρα έχουμε έντονο ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ οι μεγάλε αγορέ που καταναλώνουν στον υπόλοιπο κόσμο παραμένουν πόρτε κλειστέ για μα μας ε, επιβάλλουν κάποιο είδους ε, φυτογενομικές ε, φυτογειονομικούς περιορισμούς που είναι φραγμή χειρότερη και από τους δασμούς. Και επίσης περιορίζεται η πρόσβαση σε οποροκυπευτικά σε εκείνες τις αγορές χωρίς να υπάρχει κάποιο είδους αμοιβαιότητα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την γεωργική πολιτική ε, τα νοπά προκυπευτικά είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς και δεν καλύπτονται από τις άμεσες καταβολές. Όσον αφορά την καινούργια ΚΑΠ, τα κράτη-μέλη πρόκειται να έχουν την επιλογή να καλύψουν ε, στις ε, άμεσες ενισχύσεις αυτών των κλάδων, αλλά στην Ισπανία η κατάσταση πηγαίνει προς ε, την περιθωριοποίηση, ενώ ή τέλο πάντων προς την εξαίρεση αυτό το καθεστώς, ενώ ε, βοηθούνται ε, κάποιου είδους ε, εκμεταλλεύσεις που δεν δημιουργούν οικονομική δραστηριότητα ή απασχόληση. Και έτσι έχουμε στρεβλώσεις και δυσμενείς διακρίσεις. Όσον αφορά την έρευνα, έχουμε μια κατάσταση ρευστή, τουλάχιστον στην Ισπανία, όσον αφορά την, ε, τα, τα, τα γεωργικά προϊόντα. Οπότε και η καινοτομία δεν είναι τόσο γρήγορα εξελίξιμη όπως απαιτούν οι αγορές. Και σε αυτό το πλαίσιο, τι προτείνουμε εμείς ως ΦΕΠΕΞ Ξεκίνησε η διαδικασία της αναθεώρησης του κοινοτικού ε, καθεστώτος προκυπευτικών. Οπότε βρισκόμαστε στην, στην, στην τέλεια κατάλληλη στιγμή, ούτως ώστε να προσανατολίσουμε τις προσπάθειες προς κάποια μέτρα, τα οποία νομίζω πρέπει να εστιάζονται σε τέσσερα σημεία. Οργάνωση του κλάδου, επενδύσεις, ε, εμπορική πολιτική και έρευνα. Για την οργάνωση του κλάδου η διεύρυνση της κοινωνικής βάσης και η οικονομικής βάσης όσον αφορά τους οργανισμούς των παραγωγών προκυπευτικών είναι μια προτεραιότητα και έτσι θα διευκολύνεται η επίτευξη των ε, στόχων των επιχειρηματικών και των κλαδικών στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης αγοράς και θα ε, μεγαλώσουν οι διαστάσεις και θα επικεντρωθεί επίσης, θα, θα έχουμε συγκέντρωση προσφοράς. Γι' αυτό, αυτό το οποίο προτείνεται σε αυτή την ε, προσπάθεια μεταρρύθμισης που αρχίζει τώρα, χρειάζονται κάποια μέτρα, ούτω ώστε να έχουμε καλύτερη διαχείριση, να μην έχουμε κάποιο είδου χειραγωγήσει και να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου. Και οπότε έτσι να έχουμε κάποιε οργανώσει, κάποιου συνεταιρισμού που ενδιαφέρονται στο να καλύψουν νέα μέλη και έτσι να αυξηθεί η αξία τη ε, παραγωγή που τίθεται σε εμπορία. Από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο επίση διευκολύνεται είναι η προσβασιμότητα των νέων μελών και έτσι θα αποφύγουμε τον οικονομικό φραγμό ε, και να μην μπορεί κανεί έτσι να συμμετάσχει στο κοινωνικό κεφάλαιο. Τώρα, ως της οργάνωσης των παραγωγών, τώρα όσον αφορά τις, ε, τις, τις ε, επενδύσεις, ε, από αυτές εξαρτάται η ανταγωνιστικότητα και κατά συνέπεια η οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Τώρα, οι δράσεις οι οποίες έχουν σχέση με τη θέση σε εμπορία και το μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις ε, επενδύσεις όσον αφορά τις εκμεταλλεύσεις σαν το βασικό στοιχείο. Οπότε και εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα ενεδρεύει ο κίνδυνος του να εστιαστούν τα ε, λειτουργικά προγράμματα σε λάθος στόχους. Όσον αφορά τώρα την εμπορική πολιτική, θεωρώ δύο ε, μέτρα τα οποία θα πρέπει να τύχουν προτεραιότητας να υπάρχει αμοιβαιότητα όσον αφορά τα φυτογειονομικά και επίσης να συγκροτηθεί, να θεσπιστεί ένα καθεστώς ε, τιμή εισόδου που να είναι αποτελεσματικό. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει αμοιβιότητα όσον αφορά τα νομικά για τι εισαγωγέ. Σε μια τέτοια συγκυρία παγκοσμιοποίηση των αγορών, ε, πάρα πολλέ τρίτε χώρε απαιτούν από τα όσα εμεί εξάγουμε να τηρούν κάποια πρωτόκολλα όσον αφορά τα υγειονομικά. Κάτι το οποίο εμείς δεν το απαιτούμε από εκείνους που όταν αυτοί εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει εξομοίωση των όσων απαιτούν οι με από τους δε και Και για τα φυτογειονομικά αλλά και όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο θα, δεν θα έχουμε κάποιο είδους ε, άλλου είδους τέτοια πλήγματα στον κλάδο το δικό μας. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά τώρα το καθεστώ που διέπει εμπορική πλευρά τη εισαγωγή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είμαστε ο πρώτο εισαγωγή ε, υπολογιστικών στον κόσμο. Οπότε και οι δασμοί αντιβαλόρεμ ε, είναι πιο χαμηλοί στα σε σχέση με άλλα γεωργικά προϊόντα. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, αυτοί οι δασμοί ε, έχουν καταργηθεί μέσω εμπορικών συμφωνιών που προσυπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και συνήψε με, με τρίτες χώρες. Οπότε το να έχουμε μια τέτοια τιμολογιακή πολιτική για τις τιμές εισόδου ε, θα, πρέπει αυτό να διέπεται από αποτελεσματικότητα ούτως ώστε να σταματήσει η κατακρίμνηση των δικών μας τιμών όσον αφορά τις εισαγωγές χαμηλής τιμής. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις άμεσες σχέσεις των παραγωγών όσον αφορά την ε, έρευνα και την καινοτομία, ούτως ώστε να υπάρχει κάποιο ε, συνέχεια στις προτεραιότητες που έχουμε τάξει και αυτό θα γίνει με, με βελτίωση των ποικιλιών, με εντοπισμό και αξιοποίηση ε, των μοριακών δομών και αυτό αφορά τα, τα τα πεπόνια, τα καρπούζια, την ντομάτα και επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με κάποιες ποικιλίε όσον αφορά τα κουκούτσια ε, και επίσης κάποια άλλα τροπικά φρούτα αλλά και τα κόκκινα φρούτα, τις οργανοληπτικές ιδιότητές τους, της διατροφικής αξία και πώς θα, να δούμε πώς θα διευκολυνθεί η θέση σε εμπορία. Και με τέτοιου είδους ε, ε, μεθόδους και για τον πολλαπλασιασμό τους θα αποφύγουμε τις βασικές αρρώστιες. Και ε, όπως η Φραγκινιέλα Λοξιντεντάλη, η Μπεμίσια Ταμπάτσια, η Ακουλόψη Λικοπέρσιτζη και η Τούτα και Οπότε έτσι να αποκτήσουμε κάποιο κοινωτική νομοθεσία για την παραγωγή των προκυπευτικών και να μην έχουμε φύρα, μηδενική φύρα τέλος πάντων και έτσι να έχουμε οικολογικές καλλιέργειες θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ε, όσον αφορά το νερό, τα λιπάσματα, την ε, θέρμανση με φώτα, την, ε, τη λίπανση και το, την, τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα θερμοκήπια. να δούμε τι θα γίνει με την βιομάζα, πώς θα χρησιμοποιήσουμε ρομποτική και πληροφορική για τα για τα... En España y en la Unión Europea, orientando los recursos económicos y el esfuerzo. θερμοκήπια. Και για αυτόν τον λόγο πρέπει να δούμε πώ αυτά τα μέτρα πρόκειται να ενδυναμώσουν την παραγωγή στην Ισπανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε προ τα πρέπει να κατευθύνουμε τι προσπάθειέ μα αλλά και του οικονομικού πόρου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα. Εάν θέλετε να ακούσουμε όλους τους προσκεκλημένους μας και μετά να συζητήσουμε. Και τώρα, να λάβει το λόγο ο κύριος Ντονάτο Λαμπάτα. Ο κύριος Ντονάτο Λαμπάτα θα μας μιλήσει για τις μέλους στρατηγικές της ευκαιρίας της αγοράς. Θα μας μιλήσει για την αγορά από πλευράς των Ιταλών παραγωγών. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, επισημάνω ότι όπως ε, και εσείς γνωρίζετε η δική μας η υγεία είναι το σημαντικότερο πράγμα και δεν μπορούμε να τη διαπραγματευτούμε. Η υγεία και ε, τα τρόφιμα είναι μεγάλη σημασίας και αυτά τα δύο έχουν πολύ μεγάλο ρόλο, είναι ε, συνώνυμα της ε, ευεξίας μας, κυρίως της καλής μας ε, φυσικής ε, κατάστασης. Είναι αν θέλετε η βενζίνη του σώματός μας και ε, αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι καθαρή βενζίνη, άρα δηλαδή χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε εμείς και τα παιδιά μας. Ο τομέας των οποροκυπευτικών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και στο μέλλον θα είναι ακόμα μεγαλύτερη η σημασία του τομέα αυτού. Τα οποροκυπευτικά θα καταλάβουν τη σημασία που τους προσήκει. Εμείς ε, Είμαστε σε μια χώρα όπου αυξάνεται η ζήτηση, αυτό είναι διαμφισβήτητο, σε παγκόσμιο επίπεδο η ζήτηση τροφίμων είναι μεγαλύτερη από την προσφορά και αυτό οφείλεται όχι μόνο στην αύξηση του πληθυσμού αλλά οφείλεται και στην μεγαλύτερη κατανάλωση κατά κεφαλή. Στις αναδυόμενες χώρες ε, η ζήτηση όπως σας είπα είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά και των οποροκυπευτικών αλλά και των σιτηρών και άλλων τροφίμων που είναι καθοριστική σημασίας για την επιβίωσή τους. Άρα δηλαδή εδώ καλούμεθα να βάλουμε καινούριου στόχους στην καθημερινή ζωή. Όσον αφορά τώρα τις αλλαγές της αγοράς. Ε, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει σημαντικές αλλαγές. Ήταν ένας ε, τομέας όπου τον κύριο ρόλο έπαιζαν οι χοντρέμποροι και οι ενδιάμεση. Ε, θα θυμάστε τα παλιά καταστήματα όπου αυτά πια ήταν μικρών διαστάσεων. Αυτά όμως αντικαταστάθηκαν από την οργανωμένη διανομή η οποία και δημιούργησε και μία πόλωση στην αγορά. Υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη συγκέντρωση της ζήτησης. Πάνω από 80% των πωλήσεων λαμβάνουν χώρα μέσα από τα ε, σούπερ μάρκετ, από τα υπερκαταστήματα αυτά. Αυτό που ενδιαφέρει βέβαια είναι να υπάρχει οικονομία κλίμακας, να μπορεί να γίνει εξοικονόμηση. Ε, αυτά τα καταστήματα το καταφέρνουν και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε κάποια οικονομικά στοιχεία. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι κυρίως ε, οι μεσές επιχειρήσεις, τα φρούτα και τα απορροκυπευτικά επιτυχημένα είναι κυρίως εκείνα τα οποία περνάνε μέσα από διαδικασία νεοτερισμού και ποιοτικών χαρακτηριστικών. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες ε, είναι εξαιρετικές και σε αυτές βασίζεται κυρίως η ανάπτυξη. Αυτές οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ε, κινητήριες δυνάμεις που αξίζει τον κόπο να συγκεντρώσουν ε, χρήματα και επενδύσεις γιατί σα είπα θα μπορούσαν να οδηγήσουν προς την ανάπτυξη. Επίσης θα πρέπει να κινητοποιηθούν νέες δυνάμεις, να υπάρξουν νέα έσοδα, ε, κυρίως στον παραγωγικό τομέα. Άρα δηλαδή είναι απαραίτητο να μελετήσει κανείς την οικονομική στήριξη και τις δομές εκείνες που είναι σε θέση να ε, βοηθήσουν στην αυτοχρηματοδότηση γιατί με τον τρόπο αυτό θα προκύψουν και καλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Είναι απαραίτητο λοιπόν να μετατρέπονται οι άμεσες ενισχύσεις στην ε, γεωργία σε ε, διάρκεια ενισχύσεις γενικότερα στην γεωργία. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι μια τέτοια διαδικασία όπου θα μπορεί κανείς να αποδώσει σημασία σε αυτό το ευαίσθητο θέμα της ανάπτυξης, κυρίως στο δικό μας τον τομέα. Και αυτό που επιθυμούμε είναι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή της φοβερής κρίσης να υπάρχουν τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα επιτρέπουν την κοινωνική συνοχή, εργαλεία τα οποία θα ενθαρρύνουν χαρακτηριστικά τα οποία θα έχουν άμεση σχέση με την επιχειρηματικότητα. Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και την έρευνα. Αυτό μπορεί να δώσει κίνητρα στους νέους να ξανασκεφτούν τη Γεωργία και να στραφούν προς αυτή, να αναζητήσουν εκεί θέσεις απασχόλησης. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι επειδή εδώ βρισκόμαστε σε ένα ανώτατο επίπεδο έκφρασης μπορούν να αναλυφθούν πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν ε, στη δική μας την βελτίωση. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η εξειδικευμένη, ο ε, εξειδικευμένος τομέας. Εμείς έχουμε επιτύχει μια τέτοια εξειδίκευση, έχουμε επιτύχει την διαφοροποίηση και αυτό έχει άμεση σχέση με τις ε, τοπικές ε, καλλιέργειες. Εγώ είμαι περήφανος που είμαι Ιταλός από την Πούλια. Η δική μας η παράδοση είναι γνωστή. Έχουμε τον ήλιο, το καταπληκτικό αυτό κλίμα και επιτρέπει να προκύπτουν ειδικά χαρακτηριστικά από τα σταφύλια μέχρι τις ντομάτες. Όλα τα απορροκυπητικά έχουν ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά που οφείλονται, επαναλαμβάνω, ε, στην γεωγραφική μας θέση. Αυτά μπορούν να εξελιχθούν, μπορούν να εξυγχρονιστούν. Ε, βεβαίως, όπως σας είπα, αυτό θα πρέπει να έχει και μια οικονομική απόδοση. Η ποιότητα λοιπόν αυτή είναι μια συνταγή η οποία μας επέτρεψε να επιβιώσουμε και αυτό οφείλεται στο ότι μπορεί κανείς να αναγνωρίζει τα προϊόντα, να ε, έχει διαδικασίες χρνηλάτησης να πηγαίνει προς τα πίσω. Ο ορισμός from the farm to the table, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργασίας. Και αυτά δεν έχουν άμεση και μόνο σχέση με την, μόνο με το εμπόριο. Εμείς συνδυάζουμε την παραγωγή με την θέση σε εμπορία και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτηση στην αγορά. Το, η τυποποίηση ISO 2005 είναι ένα μοντέλο το οποίο εφαρμόζουμε ε, σε διάφορους τομείς. Όσον αφορά την διάρκεια και αυτή η διάρκεια, η βιωσιμότητα είναι μια πρόκληση για το μέλλον. Πρέπει να αποδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο θέμα αυτό. Θέλουμε και εμείς να στρέψουμε εκεί την προσοχή σας διότι η βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο το περιβάλλον και τη βιοπικιλότητα, αφορά και τα άτομα, την εργασία. Η πολιτική αυτή μας οδήγησε στο να συνεργαστούμε με τους εμπορικούς μας εταίρους, ε, με τους Biodiversity Friends ε, και αυτό οδήγησε στο να αναλυφθούν περισσότερες κοινωνικές ευθύνες. Εγώ ε, θα ήθελα να πω ότι μπορούμε να προσφέρουμε εργασία σε πάρα πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο εργασία με τη στιγμή έννοια, αλλά να τους προσφέρουμε και να τους εμπνεύσουμε σεβασμό για το περιβάλλον. Ε, αν δεν υπήρχαν βέβαια οι αγορές δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και επειδή αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των καταναλωτών οι δικοί μας οι καταναλωτές μπορούν να έχουν στο πιάτο τους φρέσκα οποροκυπευτικά κυρίως αυτή την ε, τραγική στιγμή όπου βιώνουμε μια ε, πολύ σφοδρή κρίση Τώρα λοιπόν αυτό που έχει σημασία είναι να δημιουργήσουμε απασχόληση οι χώρες BRICS ζητούν όλο και περισσότερο οποροκυπευτικά στο πιάτο τους και μπορέσαμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και εκεί και προς τη Μέση και την Αποανατολή. Έτσι λοιπόν ε, μπορεί κανείς πλέον να σκεφτεί ένα μέλλον που θα είναι πραγματικά καλύτερο. Πριν από κάποια χρόνια αυτό ήταν ένα όνειρο απατηλό, σήμερα όμως υπάρχουν τέτοιου δυνατότητες και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό καταλήξω λοιπόν στο εξή. Ε, το παλιό δίλημα που ήταν προστατευτισμός και απελευθέρωση σήμερα δεν υπάρχει πια. Η ε, πολιτική έχει την υποχρέωση πλέον να παρεμβαίνει στις αγορές με στόχο να προκύπτει μεγαλύτερη διαφάνεια και να αποφεύγονται επικίνδυνες οικονομικές κερδοσκοπίες. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει ισχυρή καθοδήγηση, μια ουσιαστική στράτευση που θα επιτρέπει όχι μόνο να αποφεύγουμε τις καταχρήσεις αλλά και οποιοδήποτε, οποιοδήποτε δόλιους στην αγορά. Κατά την άποψή μου δεν πρέπει να επιτραπεί αύξηση Τη της ε, Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στην βιοτεχνολογία, να βελτιωθεί το ανθρώπινο δυναμικό, να υπάρχει ένα δίκτυο και μέσα από αυτές τις ε, δυνατότητες ε, θα πρέπει να μπορούμε να ενισχύσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη, όπως είπε και ο συνάδελφός μου, σε συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία έχουν άμεση σχέση και με την χρήση των προϊόντων. Αυτή είναι μια, ένα στρατηγικό όραμα το οποίο συνδυάζει το όνειρο και την πράξη και έχει ως στόχο ο πρωτογενής τομέας να ε, δίδει εργασία με αρμονικό τρόπο. Όλα αυτά βέβαια έχοντας κατά νου ότι όλες οι παρεμβάσεις θα έχουν σημαντικές μακροοικονομικές επιπτώσεις. Από την ε, κατανάλωση τροφίμων μέχρι την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, όλα αυτά είναι παράγοντες πολύ μεγάλης σημασίας και για το δικό μας μέλλον και για τις επόμενες γενέσει. ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Τώρα έχουμε τον κύριο Siegfried Σόλτ, ο οποίο εκπροσωπεί τον ε, κλάδο των υπουργευτικών ή στην Γερμανία. Λέγεται Central Zentralverband Gartenbau. Καλώ ορίσατε στην ε, ακρόασή μα. Έχετε το λόγο, κύριε Σόλτ. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και επιτρέψτε μου να πω ε, και μερικά πράγματα για τα οποροκυπευτικά στη Γερμανία. Ε, σε σχέση με αυτά που ακούσαμε, εγώ θα σας παρουσιάσω μια διαφορετική εικόνα. Μια εικόνα η οποία χαρακτηρίζεται από κοινωνικές εξελίξεις αλλά επίσης ε, επηρεάζεται και από τον ανταγωνισμό έναν ανταγωνισμό ε, που ε, είναι έντονος σε αυτόν τον τομέα η προσαρμογή, ο προσανατολισμός προς την αγορά, αυτό πάντα για μας ανέκαθεν ήταν καθοριστική σημασία και έχω τέσσερα σημεία που θέλω να σας αναφέρω. Καταρχήν μια γενική εικόνα για την ποικιλομορφία στην αγορά, στη Γερμανία, κατόπιν ε, κινδύνους και θα ήθελα ε, επίσης να σας παρουσιάσω και μια προοπτική που ακριβώς βλέπουμε να υπάρχουν προκλήσεις και στο τέλος θα κάνω κάποιες ε, συνοπτικές παρατηρήσεις. Και νομίζω αφορά τα συμπεράσματα τουλάχιστον, συμφωνώ με τους ε, συναδέλφους μου. Ε, θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Βλέπετε ότι τα οποροκυπευτικά είναι καθοριστική σημασίας. Ε, έχουμε όμως και πολλά άλλα διακοσμητικά φυτά και με όλα αυτά καλύπτουμε ένα μεγάλο φάσμα, μια μεγάλη βεντάλια προϊόντων. Θεωρώ λοιπόν ότι στο λιανικό εμπόριο και στην παροχή υπηρεσιών υπάρχουν άμεσες διασυνδέσεις όσον αφορά την παραγωγή. Και όλα αυτά έχουν σχέση με την παραγωγή, το λιανικό εμπόριο, αλλά ακόμα και τα οπορικυπευτικά, τα διακοσμητικά αυτά που καλλιεργούνται για τα νεκροταφεία και αυτά είναι ένα σημαντικό τομέα. Και βλέπετε λοιπόν ότι ε, όπως σας είπα, η δική μας η καλλιέργεια είναι καθοριστική σημασία και για την καλλιέργεια φυτών. Τον Απρίλιο αυτού του έτους ε, το Υπουργείο μας ε, παρουσίασε αυτή τη μελέτη που βλέπετε και στη διαφάνεια ε, που είναι από ένα Ινστιτούτο στο Braunschweig. Αυτή λοιπόν η μελέτη δείχνει ότι στο κέντρο Έχουμε την ε, ε, πρωτογενή παραγωγή με φυτά, λουλούδια, οποροκυπευτικά και γύρω-γύρω έχουμε πάρα πολλές άλλες διεργασίες που κατατάσσονται στην οποροκυπευτική και αυτό πολλοί το αγνοούν. Δηλαδή, γίνεται καλλιέργεια οποροκυπευτικών σε μεγάλες εκτάσεις, πολλοί όμως ξεχνάνε ότι πίσω από αυτό υπάρχουν διάφορες υποδομές. Αυτό λοιπόν φαίνεται εδώ στη διαφάνεια, στη μελέτη που έκανε το Υπουργείο και βλέπουμε ότι παίζουν ρόλο πολλά πράγματα όπως οι διαβουλεύσεις για την εκπαίδευση αλλά και γενικότερα στην Αγγλία ας πούμε αν δεν υπήρχαν αυτοί οι φοβεροί κήποι της Αγγλίας ποιος θα πήγαινε τουρίστα στην Αγγλία έλατε όσον αφορά τη σημασία αυτού του τομέα Βλέπετε εδώ ε, κάποια παραδείγματα που αφορούν την παραγωγή. 1,8 δις ευρώ δαπανήθηκαν για απορροκυπευτικά. 400 εκατομμύρια για τα φρούτα, ε, κάποια άλλα 400 εκατομμύρια για τα διακοσμητικά φυτά. Βλέπετε δηλαδή ότι μιλάμε για περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ που εστιάζονται στην παραγωγή. Αν όμως δούμε λιγάκι και το εμπόριο, θέλω να σας καταστήσω σαφές ότι όσον αφορά την παραγωγή και τη διασύνδεσή της με την παροχή υπηρεσιών, διαπιστώνουμε ότι αυτά τα 5 δισεκατομμύρια όπου περιλαμβάνονται και τα κονδύλια που αφορούν στην καλλιέργεια φυτών για τα νεκροταφεία. Αυτό λοιπόν είναι το ποσό που αφορά το σύνολο των οποροκυπευτικών, όπου προστίθενται και διάφορα άλλα επιμέρους ποσά και καταλήγουμε στα 16 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό και αν συμπεριλάβουμε και την μεταποίηση στον ε, τομέα της ε, χοντρικής πριν και μετά την πώληση, Εάν λοιπόν τα προσθέσουμε και αυτά, καταλήγουμε τελικά σε 78 δις ευρώ, τα οποία 78 δις ευρώ αφορούν αλλά και περιστρέφονται γύρω από ε, γενικότερα την ευρία έννοια των απορροκυπευτικών. Και τώρα θα πω και δύο άλλα πράγματα σχετικά με τις εξελίξεις. Αν δούμε λιγάκι τη ζήτηση και τη δημογραφική εξέλιξη θα διαπιστώσουμε ότι το σύνολο της ζήτησης για τα δικά μας τα προϊόντα είναι υψηλή και αυξάνεται περισσότερο η ζήτηση αυτή. Έχουμε κάνει διάφορες μελέτες και διαπιστώνουμε ότι οι δημογραφικές αλλαγές αλλάζουν και τις απαιτήσει, παραδείγματος χάρη μια σημαντική απέτηση που εμφανίζεται πλέον είναι η βιωσιμότητα. Όμως εκείνο που επίσης ενδιαφέρει είναι ότι υπάρχει μια τάση εντοπιότητας να δίδεται σημασία στα τοπικά προϊόντα. Παίζουν ρόλο αυτά ακόμα και στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου η συνειδητοποίηση περί ποιότητας. Αυτή είναι όλο και μεγαλύτερη. Στον τομέα αυτό αναλαμβάνουμε πολλές προσπάθειες. Έχουμε μια γενιά που θα δώσει όλο και περισσότερη σημασία στη διατροφή αλλά και στην περιραίουσα, στα όλα τα συμπαρομαρτούντα. Ε, γι' αυτό λοιπόν όπως ε, σας είπα ε, ασχολούμεθα και με άλλους τομείς, ε, υποτομείς, την ανθοκομία μεταξύ άλλων αυτό που θέλω να τονίσω και αναφέρθηκε αυτό ε, στην τελευταία παρέμβαση, αυτό που θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο είναι ότι θέλουμε να έχουμε ικανούς εργαζόμενους. Αυτό ισχύει ε, και στην παροχή υπηρεσιών και στην παραγωγή. Τα απορροκυπευτικά, η ανθοκομεία ε, με τον εκμηχανισμό διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι ο ανταγωνισμός. Εδώ διαπιστώνουμε ότι ε, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη προσφορά. Βλέπουμε την συγκέντρωση σε discounters και κατόπιν του είναι σαφές ε, ότι επικρατεί μεγάλος ε, ανταγωνισμός και αν ε, προσθέσουμε και τις ε, ε, συνθήκες τις κλιματικές, καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Θα ήθελα να αναφέρω το θέμα των διακοσμητικών φυτών. Σε 10 χρόνια διαπιστώθηκε μείωση της παραγωγής της τάξης του 22%. Εδώ διαπιστώνουμε μια μεγάλη αλλαγή. Πλέον υπάρχει συγκέντρωση στην παραγωγή. Μας ενδιαφέρει και περισσότερο η ε, παραγωγή με χαμηλότερο κόστος. Εξορθολογισμός δηλαδή. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχουν ε, πολλές ευκαιρίες και για μικρές επιχειρήσεις, όχι μόνο σε εξειδικευμένες αγορές, αλλά σας είπα προηγουμένως ότι η εντοπιότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό και περίπου το 35% των προϊόντων τοποθετείται στην αγορά μέσα από ενός παραγωγών. Το 35%, το 65% ακολουθεί ε, άλλους δρόμους. Αυτά δεν πρέπει να τα παραγνωρίζουμε στο βαθμό που θέλουμε να έχουμε μια τέτοια πολιτική που θα βοηθάει και τον παραγωγό. Επαναλαμβάνω, ε, Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προβάλλουμε το στοιχείο της εντοπιότητας, της περιφερειακής ανάπτυξης. Για να δούμε τώρα λιγάκι τι μπορείτε να κάνετε εσείς, τι περιμένουμε από την Ευρώπη. Περιμένουμε τη στήριξη της ε, βιωσιμότητας, να υπάρχει επάρκεια πόρων ε, στο πλαίσιο της, ε, κυρίως αναφορά τον εφοδιασμό με ενέργεια. Και ένα άλλο παράδειγμα που θέλω να αναφέρω είναι ότι στον τομέα των δικτών και των κενών που καταγράφουν οι δείκτες Υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις, πρέπει λοιπόν να υπάρξει προγραμματισμός έτσι ώστε να καταλήξουμε συμπεράσματα και αποτελέσματα που θα βοηθήσει όλους. Ε, έρευνα και ανάπτυξη, το έθιξε ο συνάδελφος, πράγματι και εμείς αναγνωρίζουμε ότι στον τομέα αυτό ε, χρειαζόμαστε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα καινοτομίας. Ε, εμείς στη Γερμανία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα αποτελέσματα. Η πρόθεση των πωλήσεων για όλους, για μας αυτό είναι καθοριστική σημασία. Πρέπει να μεριμνήσουμε, γιατί πράγματι οφείλουμε να ενισχύσουμε τις ενώσεις παραγωγών, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατ' ουσίαν θα πρέπει παράλληλα να δημιουργήσουμε και άλλα στοιχεία που να βοηθήσουν παρεμφερείς επιχειρήσεις. Όπως σα είπα η διάθεση των πωλήσεων στον δεύτερο πυλώνα ενίσχυση της εντοπιότητας. Αυτό σημαίνει και ενίσχυση της διάθεσης των ε, πωλήσεων. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω εσείς ε, ε, θα επιληφθείτε του θέματος αυτού. Η γραφειοκρατία είναι κάτι που απασχολεί πάρα δικούς μας τους ε, μικροκαλλιεργητές. Και ανακεφαλαιώνω, η οικονομική σημασία των οπεροκυπευτικών και της ανθοκομείας γενικότερα του τομέα πολύ συχνά υποτιμάται. Ε, εμείς καλύπτουμε βέβαια το 1% της συνολικής ε, καλλιεργήσιμης έκπτωσης στη Γεωργία. Η υγιής διατροφή πρέπει να συνεχίσει να στηρίζεται και αυτό που ενδιαφέρει είναι κυρίως οι νέοι να τρέφονται σωστά. Ευελικτή ευημερία λοιπόν και ευεξία. α μην ξεχνάμε και την περιραίουσα ατμόσφαιρα και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να επισημάνουμε λιγάκι και το θέμα της ανθοκομίας γιατί και η ανθοκομία έχει πολιτιστική αξία και όταν θα τοποθετηθείτε επί του ΦΠΑ και του πρώτου παρατήματος παρακαλώ να καταστήσετε σαφές ότι τα λουλούδια γενικότερα είναι ένα πολιτιστικό στοιχείο το οποίο όμως μπορεί να το και κάτω από το πρίσμα της υπεραξίας καθαρές πόλεις, ε, καθαρή ατμόσφαιρα. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία εμείς προάγουμε και βλέπετε εδώ ε, κάποια στοιχεία που, ε, τα οποία εντάσσουμε στο δικό μας το σύστημα ενημέρωσης, το Hortgate. Προηγουμένως ακούστηκε ότι το πρόβλημα είναι τα επιστημονικά δεδομένα να τα μετατρέψουμε στην πράξη. Να, ειδού, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα, εδώ και 10 χρόνια, όπου για τα απορροκυπευτικά, για τα φυτά και για άλλους τομείς έχουμε πληροφορίες που διοχετεύονται άμεσα στους ε, παραγωγούς και επ' αυτού συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι επιστήμονες του τομέα. Κυρίες και κύριοι, η βιώσιμη παραγωγή ε, με μέρημνα στην ενέργεια. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Ε, νομίζω ο δικός μας ο τομέας εμφανίζεται διαφοροποιημένος. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ο Πρόεδρος. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτριά μας να κάνει τι ε, να δευτερολογήσει τέλο πάντων τις καταληκτικές της παρατηρήσεις και να ακολουθήσουν τυχόν ερωταπαντήσεις. Οπότε, ο πρώτος ο οποίος τώρα έχει ζητήσει το λόγο είναι η κυρία Γκαρθία. Κυρία Γκαρθία, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τέσσερις προσκεκλημένους, τους εισηγητές μας, νομίζω ότι πρέπει να του ευχαριστήσουμε που ήρθαν εδώ να μας μιλήσουν για έναν τόσο σημαντικό κλάδο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ιδιαίτερα και για την δική μου χώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε στην κεντρική Ισπανία, παντού, παντού, βορρά, νότο, ανατολή, δύση και στη Γαλλική. Πάρα πολύ σημαντικός κλάδος. Ε, λυπάμαι που δεν μπόρεσα να είμαι εδώ και να ακούσω τον πρώτο εισηγητή, αλλά ήμουν στην Επιτροπή Αναφορών. Εκεί είχαμε έναν αναφέροντα που μιλούσε για το Δέλτα του Εύρου. Και εκεί έχουμε κάποιους συνεταιρισμούς και εκεί έχουμε παραγωγή προκυπευτικών και δυστυχώς ήθελα να σας πω ότι υπήρξε έντονη επίκριση ε, από τους αναφέροντες για τον τρόπο που ποτίζεται το δέλτα του ευρώ η λεκάνη τέλο πάντων αυτή ε, του, του, ποταμού ευρώ Πάντως, έχουμε τώρα νέους ορίζοντες που ξανοίγονται με αυτή τη νέα έκθεση που θα ζητήσω αμέσω στους μήνες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα διαχειριστούμε την κρίση. Απόσυρση, συγκομιδή, ενημέρωση, ασφάλειες, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση με τις αποσύρσεις, πώς θα διαχειριστούμε έτσι την κρίση. Με τις αντισταθμίσεις θα πρέπει να δούμε πώς θα ε, διαχειριστούμε την αγορά και πώς θα συνδέσουμε την απόσυρση με τις ενισχύσεις για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Στην Ισπανία αλλά και στην ε, Γαλλία πρόσφατα είχαμε και κάποια συνεννόηση που ενσωματώθηκε σε κάποια συμφωνία. Ζητήθηκε μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά. Ζητήθηκε αναβάθμιση των οργανώσεων παραγωγών. Νέο νομοθετικό πλαίσιο ανταγωνισμό, γιατί ξέρετε στην Ισπανία έχουν πρόβλημα την ε, ε, το σχετικό φορέα, τον κρατικό. Υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές εισόδου των εισαγωγών. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ αυτή την κατεύθυνση. Με το να εξεύρουμε έναν πιο αποτελεσματικό, πιο δόκιμο μηχανισμό. Έτσι, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα βασικά προβλήματα και τα φαινόμενα απάτης που είχαν αναφυεί στο παρελθόν. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη από τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Και έτσι να έχουμε καινούριο καθεστώς τιμών εισόδου και αυτά όλα να ενσωματωθούν σε κανονισμού. Τώρα, να αφορά την προστασία του περιβάλλοντο, την καταπολέμηση των ε, ασθενειών, θα πρέπει να έχουν πιο ευέλικτη νομοθεσία. Έχουμε τώρα και τι πρόσφατε αυτέ περικοπέ. Έχουμε τους περιορισμούς όσον αφορά τις δραστικές ουσίες για τις φυτογενομικές, για τις ασθένειες τέλος πάντων. Όλα αυτά και έχουν καταστήσει ακόμη πιο ευάλωτο τον τομέα. Άρα πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Γιατί έχουμε βρεθεί τώρα πάρα πολύ ακάλυπτοι. Εδώ έχει ασχοληθεί και η παρακαθήμενη, συνάδελφος, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να δούμε για τα φυτογενομικά και τα σχετικά προβλήματα. Θα πρέπει να είναι πιο ευαίσθητη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αμοιβαιότητα για αυτούς τους φραγμούς, τους περιορισμούς, τους φυτογενομικούς που επιβάλλουν τρίτες χώρες όπως Βραζιλία ή ΙΠΑ. Σπάνια, σπάνια δεν χρειάζεται να διαμαρτυρηθούμε ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια περίοδο συγκεκριμένη εμπορία για τα προβλήματα από τις τρίτες αυτές χώρες. Ήδη τώρα έχουμε προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά για την παραγωγή που προέρχεται από τρίτες χώρες όπως είναι τη Φραγική Δημοκρατία και άλλα προβλήματα που ανακύπτουν. Άρα θα πρέπει να επαγρυπνούμε για το τι μπαίνει από τα σύνορα, τι εισαγωγέ γίνονται. Άρα θα πρέπει να ζοριστούμε από την έκφραση για να προστατευτούμε από τις εισαγωγές των χωρών. Πολλές φορές ε, μπαίνουν και άρρωστα φυτά οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Ε, μην καταντήσουμε σαν το φίδι το οποίο κυνηγάει την ώρα του γύρω γύρω και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Χωρίς να βρίσκουμε τη λύση λοιπόν. Έχουμε το σχετικό έγγραφο ε, για την νέα αγορά, για την κοινή οργάνωση αγοράς μάλλον, για την νέα αγορά. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις διεθνείς συμφωνίες. Υπάρχει τώρα ε, η διαδρομή των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με, την, με τις γεωγραφικές ενδείξεις, με την ονομασία προέλευσης και θα πρέπει επίσης να δούμε το θέμα της αμοιβαιότητας με τις τρίτες χώρες. Θα είναι πολύ σημαντική η συμφωνία που θα συμπήξουμε, που θα κλείσουμε με τις ΙΠΑ. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις ενδείξεις των, ε, γεωγραφικών, ε, των αγροτικών προϊόντων, κάτι τόσο σημαντικό για την Ένωση. Ο Πρόεδρος. Και τώρα έχει το λόγο η κυρία Αγίουσου. <coughs> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Α, συγγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα καλά ότι έδωσα το λόγο σε μένα. Να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους εισηγητές για τόσο μας εξήγησαν που, για την περιγραφή της κατάστασης του κλάδου των προγευευτικών στη χώρα του καθενός. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια για αυτή την έκθεση και ε, θα δούμε πώς θα ρυθμιστεί η καινούργια κοινή οργάνωση αγοράς για το προγευευτικά. Όλα όσα μας είπατε κύριοι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Να μην επαναλάβω αυτά που είπε η Εστήρα εδώ εκ δεξιών μου, αλλά όσον αφορά την αμοιβαιότητα για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τα φυτογειονομικά, ναι, και εδώ θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγώ δουλεύω και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, την Κοινοβουλευτική και συζητούμε πολύ συχνά το πόσο βλάπτουν οι παραγωγοί τομείς από τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα. Θα πρέπει κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συνέπειες, ξέρετε, αυτής τη κατάστασης είναι τεράστιες, ήταν πολύ μακριά. Δεν είναι θέμα της δόσης, τις ελάχιστες δόσεις κλπ. Για μένα το πρόβλημα αυτό είναι από τα πιο σημαντικά που έχουμε αντιμετωπίσουμε. Αυτό αφορά όλο τον Νότο. Άλλωστε άλλε ασθένειε και άλλα έντομα έχουμε στο Νότο. Στο Βορρά επίση, ε, απαγορεύονται κάποια προϊόντα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και που τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ την παραγωγή. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Άλλο θέμα σημαντικό είναι το καθεστώς που διέπει τις τιμές εισόδου. Και όσον αφορά την έρευνα, έχω ασχοληθεί με την γεωρική έρευνα 20 χρόνια. Ξέρω τον κλάδο. Έχω πάει σε πάρα πολλά θερμοκήπια. Θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για τους ερευνητές, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία εύρυθμη με τα ερευνητικά κέντρα στη χώρα του καθενός και αν κατακλείδη υπάρχει κάτι άλλο το οποίο αναφέρθηκε. Το θέμα των ενισχύσεων ανά εκτάριο. Στη χώρα μου λένε ότι μόνο οι μεταποιητές λαμβάνουν άμεση ενίσχυση. Τώρα θέλουμε να μας πούνε οι παραγωγοί των προκυπευτικών. Τι προτιμάνε. Την ενίσχυση ανακτάριο. Γιατί πολλές φορές αυτό που παίρνουν είναι γελίο, είναι φραγκοδίφραγκο. Ή μήπως το προτιμούσαν κάποιους ε, λειτουργικά επιχειρησιακά ταμεία. όπως πάει τώρα η ΚΑΠ, δεν θα έχουμε τελικά την σημαντική κοινή οργάνωση αγοράς για το προκυπευτικά. Πέστε μας τη γνώμη σας. Καλά και πέραν του θέματος της ενίσχυσης ανεκτάδη. Θα πρέπει να μπορούν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το προκυπευτικά να ε, μπορούν να είναι σύγχρονες, να εξυγχρονίζονται και να είναι ανταγωνιστικές. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα. Κυρία Ρόντουστ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τέσσερις ε, ομιλητές. Εγώ πραγματικά πήρα πολύ σοβαρά αυτά που μας είπαν με την έννοια ότι η έκανε μία παρουσίαση αρκετά αρνητική. Ο τομέας αυτός πραγματικά έχει δυνατότητες. Πρέπει να προωθήσουμε τα συμφέροντά τους. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Τελικά όμως βλέπουμε ότι πρόκειται για έναν τομέα με προοπτικές και σας ευχαριστώ πολύ γιατί αναφερθήκατε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και στις οποίες πρέπει εμείς να πάρουμε σοβαρά υπόψη μας. Άκουσα πολύ προσεκτικά από έναν από εσάς ότι το θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης και είναι πολύ σημαντικό. Έχετε δίκιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πανεπιστημιακά ιδρύματα με προτάσεις καινοτομίας και ιδέες στην έρευνα. Και θα πρέπει εδώ βεβαίως να υπάρξει σύνδεσμος μεταξύ του δικού σας τομέας και της νέας τεχνολογίας, της έρευνας. Παραδείγματο χάρη, στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου άκουσα μια πολύ καινούρια ιδέα όσον αφορά την ίδρευση, όσον αφορά νέες δυνατότητες ε, παροχής ε, νερού για τις καλλιέργειες. Πώς βλέπετε εσείς ε, αυτές τις ιδέες, τι έχετε να πείτε, τι είναι οι ανάγκες του τομέα. Επίσης, όσον αφορά τις υδατοκαλλιέργειες στον τομέα της αλληλείας, ιδιαίτερα για υδατοκαλλιέργειες σε γλυκά νερά. Ξέρουμε ότι υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης αυτών των υδάτων και για κάποιες καλλιέργειες και το νερό αυτό το οποίο ξαναχρησιμοποιείται και ξαναδίνεται κατόπιν παρέχεται στην ε, καλλιέργεια ε, αυτή από την ε, παραγωγή δηλαδή φυτών στην ηχθειοκαλλιέργεια. Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με μικρές μονάδες παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν αυτό το νερό μα είπατε όλοι ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο τοπικός χαρακτήρας των προϊόντων, οι μικρές περιφερειακές καλλιέργειες, οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Και από ό,τι φαίνεται πρόκειται για ένα κλειστό κύκλωμα χωρίς την ε, χρησιμοποίηση συγκεκριμένων ε, ουσιών που μολύνουν το νερό, χωρίς ε, τον περιορισμό της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα και με πολύ πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές. Μπορούμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Εγώ παρακολούθησα δύο συγκεκριμένες ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν αυτές τις πρακτικές, αυτές τις νέες τεχνικές. Στη μία περίπτωση ήταν ε, λαχανικά και στις άλλες ε, ήταν ε, η συμμετοχή ύδατος σε υδατοκαλλιέργειες και ηχθειοκαλλιέργειες. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Έχετε το λόγο. Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για αυτές τις ε, παρεμβάσεις. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Βεβαίως ε, υπάρχουν και κάποιες διαφορές που άκουσα. Ας πούμε στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε, έχουν κλείσει κάποιες επιχειρήσεις στον τομέα των οπορικπευτικών. Σε άλλες πάλι ακούσαμε για ενός παραγωγών ότι αυτή είναι η καλή λύση, η λύση του μέλλοντος. Βέβαια πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε να μην κυριαρχήσουν τελικά οι ενώσεις παραγωγών. Γιατί οι επιχειρήσεις που δεν δεν θα εντάσσονται σε ενό παραγωγών, αυτές θα υποστούν στρέβλωση τη αγορά. Αυτό που ενδιαφέρει λοιπόν να υπάρξει κάποια ισορροπία. Και αυτό που έχει επίση ενδιαφέρον είναι ε, το ότι τα οποροκυπευτικά μαζί με τα διακοσμητικά φυτά ε, είναι καθοριστική σημασία για την κοινωνία, Εκεί υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επαφή με πολίτες από τη γενικότερα ας πούμε στη Γεωργία γιατί αυτή η μορφή Γεωργίας επιτρέπει την καθημερινή επαφή. Θεωρώ λοιπόν στον δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την καλλιέργεια οποροκυπευτικών δηλαδή να υπάρχουν ε, συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτό που θα με ενδιέφερε είναι το εξή. Ε, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο πακέτο για τους σπόρους, θέλαμε να γνωρίζουμε ε, τι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ε, σε σχέση ε, με την καλλιέργεια όποροκυπευτικών. Και όσον αφορά την διαχείριση της υγείας και γενικότερα των ασθενειών, τα ζυζανιοκτώνα πώς ακριβώς ε, τα εντάσσεται, κυρίως αυτά που αφορούν ασθένειες ε, καραντίνας, που οδηγούν σε καραντίνα. Υπάρχουν μέτρα για να καλυπτώμεθα. Και ποια είναι τα μέτρα εκείνα έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μην καταστρέφονται, να μην απειλούνται με οικονομική καταστροφή διότι όσο νωρίτερα ε, αναφέρονται τα ζενοκτώνα που αφορούν ασθένειες καραντίνας, τόσο καλύτερα. Τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος ε, τελικά να προκύψει συνολική ζημιά για τον τομέα. Εμένα λοιπόν με ενδιαφέρει να μας πείτε εσείς πώς ακριβώς βλέπετε το θέμα. Ο πρόεδρος. Κύριος Χάσλεκ. τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις έχω και φυσικά θα μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που άκουσα όσον αφορά την γραφειοκρατία. Εμείς σας υποσχόμαστε με τη νέα αναθεώρηση βελτίωση. Πώς το βλέπετε εσείς, ποιες είναι οι συγκεκριμένες ε, ε, απαιτήσεις σας όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τη καλύτερες, ε, πιο φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Εγώ εδώ ακούγοντας τον Βρετανό ομιλητή άκουσα κάποια κριτική, ιδιαίτερα όσον αφορά την αποχώρευση των ουσιών αυτών που βλάπτουν τις μέλισσες. Το θέμα της χρήσης χημικών ουσιών. Ναι, βέβαια, υπάρχουν πολλές παραβιάσεις των ανώτατων ορίων όσον αφορά την περιεκτικότητα κάποιων ε, τοξικών ουσιών. Αυτό καταλαβαίνετε ότι πάντα με προβληματίζει. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Από τη μία έχουμε τους παραγωγούς, ε, την απόδοση των καλλιεργειών. Από την άλλη πρέπει να είμαστε ε, ευαίσθητοι στην προστασία του περιβάλλοντος και βεβαίως πρέπει αυτές οι τοξικές ουσίες να μειωθούν. Όσον αφορά την ανθοκομία και τις τρίτες χώρες, τις εισαγωγές, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις συνθήκες εργασίας παραγωγής στις τρίτες χώρες με αυτές που ισχύουν στην Ευρώπη. Το ανθρώπινο δυναμικό, το εργατικό δυναμικό εκεί, θα το πω προσεκτικά, βασίζεται σε άλλου είδου συνθήκε εργασία σε εκμετάλλευση και μετά αυτά τα προϊόντα εισάγονται στην Ευρώπη. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό έτσι ώστε να μην την πληρώνουν πάντα οι εργαζόμενοι. Να βρούμε μια έξυπνη λύση. Bardzo proszę ostatni głos dyskusji pan poseł <clears throat> Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους για όσα είπανε και εγώ συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που ακούσαμε ακριβώς όπως τα είπαν εδώ και οι Ισπανίδες ε, συνάδελφοι. Σύμφωνα και με εκείνε. Αλλά θέλω να σα πω κάτι άλλο, κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορούμε να μιλούμε για το μέλλον του κλάδου γενικά όταν δεν τον πρεκοδοτούμε για να του εγγυόμεθα το μέλλον να υπάρχει επομένω η προκοδότηση, να υπάρχει το νομικό πλαίσιο και επίσης αυτά που συμφωνήσαμε να τα τηρούμε. Άλλο η θεωρία, άλλο τα μεγάλα λόγια και άλλο το τι κάνουμε στην πράξη. Ε, στην πράξη κάθε μέρα, γιατί έχουν στριμωχτεί πάρα πολλοί παραγωγοί και βλέπουν μελανό το μέλλον, με μελανά χρώματα. Οπότε, ξέρετε, τα προεκυπευτικά είναι πάρα πολύ σημαντικά για τα Κανάρια νησιά. Σήμερα έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ ο κλάδος και άρα χρειάζονται μέτρα τα οποία θα φρενάρουν αυτή την επικίνδυνη κατηφορική πορεία που έχει πάρει. Μιλάμε για αμοιβαιότητα. Ωραία. Αλλά πέραν αυτό έχουμε κάποιες ποσοστώσεις. Εντάξει. Έχουμε μέσα αναφοράς. Επίσης που έχει γίνει προσπάθεια να βελτιωθούν αλλάζοντας το σύστημα. Αλλά μέχρι ποιο σημείο αυτό το σύστημα έχει εγγύησεις ε, της του του, της συμμόρφωσης προς αυτό, θα πρέπει τα ίδια τα θεσμικά όργανα να παρέχουν εγγύησεις στήριξης, της συμμόρφωσης προς το σύστημα. Επαναλαμβάνω, γενικά ακούμε πολλές δηλώσεις, αλλά συγκεκριμένα για τα καθημερινά ζητήματα δεν φροντίζουμε να τηρούνται αυτά τα οποία εμείς οι ίδιοι αποφασίζουμε. Αλλιώς, έτσι, αν δεν κάνουμε κάτι, δεν έχει μέλλον ο κλάδος. Κάτι να κάνουμε για να προστατεύσουμε τη δική μας παραγωγή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, οι προσκεκλημένοι μας, αν θέλουν, να δώσουν κάποιες σύντομες απαντήσεις προς τις ερωτήσεις. με την ίδια σειρά με την οποία κάνατε την εισήγηση. Ε, ναι, να σας πω πρώτα πρώτα ε, σε εσάς ε, συμπατριώτησα κυρία Αγιούσο που αναφερθήκατε στα λειτουργικά επιχειρησιακά ταμεία, τις σχετικές ενισχύσεις, τις άμεσες ενισχύσεις. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ απλή η απάντηση. Ναι, και το ένα και το άλλο. Όπως ε, είπατε, γιατί τα λειτουργικά επιχειρησιακά προγράμματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις οργανώσεις των παραγωγών και όπως ανέφερα τον έλαβα το λόγο αυτά έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις και οι επενδύσεις βοηθούν το να είμαστε ανταγωνιστικοί και να, ε, και να έχουμε καινοτομία. Με τη νέα κοινωνική πολιτική θα καλύπτονται από τις άμεσες ενισχύσεις και τα προεκυβευτικά. Όμως, το πρόβλημα είναι ότι μια που αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα, τι θα γίνει εάν ε, κάποιο προκυπευτικό, κάποιο συγκεκριμένο προϊόν δεν την χάνει ενίσχυση στην Ισπανία, αλλά την χάνει ενίσχυση σε άλλη χώρα. Αυτό θα οδηγήσει σε του διαγωνισμού. Αυτό θέλω να σας πω μόνο. Δεν θα ξεκινήσω τα σχόλιά μου για αυτά που ακούστηκαν για την υδατοκαλλιέργεια και τη χρησιμοποίηση των υδάτων αυτών για άρδευση. Αυτό είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Όσον αφορά τα σχόλια που κάνατε, σαφώς και η παραγωγή μειώνεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο και φυσικά και η χρήση των ε, τοξικών αυτών ουσιών στα ζυζανιοκτώνα και σε άλλες ε, ουσίες που χρησιμοποιούνται μειώνεται και είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Φυσικά και είναι μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι να μπορούμε να αποδείξουμε τον τοπικό χαρακτήρα των προϊόντων. Αυτό είναι σημαντικό και για την αλυσίδα ε, διατροφής και για την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και πολύ συγκεκριμένα για την ανάπτυξη των περιφερειών μας. Και το πιο σημαντικό μήνυμα που έχω να σας δώσω σήμερα είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τομέας μας ο οποίος πολλές φορές δεν είναι γνωστός, δεν είναι γνωστή η σημασία του και η αξία του. Πρέπει να συνεχίσουμε να τρώμε λαχανικά και φρούτα, μία μικρή αύξηση της κατανάλωσης οποροκυπευτικών προϊόντων θα βοηθήσει και τους παραγωγούς αλλά και στην βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων καταναλωτών. Αυτό είναι το μήνυμά μου, είναι πολύ απλό. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι συνάδελφοι έθιξαν περίπου τα ίδια προβλήματα και πρώτα περίπου τις ίδιες λύσεις. Δηλαδή, σαν να είχαμε μιλήσει εκ των προτέρων μεταξύ μας για τα προβλήματα. Και θα ήθελα να απαντήσω σύντομα στην πολύ καλή κυρία από την Ισπανία για το θέμα των επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι απαραίτητο να δίδουμε ενισχύσει, αλλά όχι ε, χωρίς καμία διάκριση ενισχύσει, επειδή βρέχει, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό είναι καθοριστική σημασία κατά την άποψή μου να υπάρχει ένα εργαλείο ένα είδος ε, τράπεζας, αλλά όχι εμπορική τράπεζα, μία ε, τράπεζα ενίσχυσης. Ε, νομίζω αυτό το θέλουμε όλοι στην Ευρώπη. Να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στην Ευρώπη. Μία τράπεζα ενισχύσεων που θα καταθέτει ε, τις ε, επιδοτήσεις όχι τυχαία αλλά πολύ συγκεκριμένα. Ίσως ε, αυτά που λέω να είναι πολύ οικονομικά και πολύ στοχευμένα σε θέματα οικονομίας, αλλά ξέρετε στην Ιταλία, όπως και γενικά στον νότο της Ευρώπης, ε, ο μεταποιητικός τομέας αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες και τώρα βρισκόμαστε σε μια νέα φάση. Η Γεωργία προσφέρει νέες δυνατότητες, επενδύσεις που γενικεύονται και αυτό ε, νομίζω μπορεί να φέρει την ευημερία, όχι μόνο την ατομική ευεξία, αλλά μπορεί, αν θέλετε, να φέρει και την κοινωνική ευημερία. Και κάτι άλλο που θέλω να πω, γιατί ακούσαμε πάρα πολλές και καλές ε, επεμβάσεις, αλλά ο χρόνος δεν φτάνει, είναι ο τύρανός μας. Κοιτάξτε, έχω κατά νου μια συγκεκριμένη ιδέα. Ένα κόσμο έχουμε, δεν έχουμε άλλον και αυτόν καλούμεθα να τον προστατεύσουμε. Ε, βλέπω λοιπόν ότι έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο τουλάχιστον όσον αφορά τα τρόφιμα και με τα χέρια μας μπορούμε να προστατεύσουμε ή να καταστρέψουμε αυτό τον πλανήτη. Αυτό που οφείλουμε να ζητήσουμε είναι καθαρές μορφές ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές, ηλιακή ενέργεια ή αιωλική ενέργεια που δεν ρηπαίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ που οργανώσατε αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ο κύριος ε, Σόλτς. Εγώ λοιπόν ε, θα ήθελα να ξεκινήσω ε, σε αυτά που ρώτησε η Ταλίδα ε, η συνάδελφός μας σχετικά με τα μέτρα φυτοϊγειονομικής προστασίας. Κοιτάξτε, από την Ρωσία βλέπουμε ότι επιβάλλονται εμπορικοί φραγμοί που δεν είναι απαραίτητοι. Στους ε, Ισπανούς συναδέλφους θέλω να πω ότι η αντιπαράθεση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, υπάρχει σε θέματα εγκρίσεων αυτό μπορούμε να το στηρίξουμε, δηλαδή ε, να υπάρχει κάποια ενίσχυση στον τομέα των, φυτών στον ανθοκομικό τομέα έτσι ώστε και να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους ανθρώπους. Και επίσης ε, θέλω να απαντήσω και στον κύριο Χόισλινγκ. Πράγματι νομίζω μπορούμε να απαντήσουμε ανεπιφύλακτα ναι ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση ως ε, προς τη μείωση των κινδύνων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μειώνονται απαραίτητα και οι ποσότητες. Όλα εξαρτώνται από την δηλητηριώδη μορφή, από την χρήση και εδώ και πολλά χρόνια σε στρογγυλές τράπεζες προσπαθούμε να καλύψουμε κάποια κενά. Νομίζω λοιπόν ότι ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο αν μπορείτε να μας βοηθήσετε, κυρίως αφορά τις ε, μικροκαλλιέργειες. Ε, αυτά που είπατε για το σύστημα aquaponic, τον συνδυασμό υδατοκαλλιέργειας με καλλιέργεια φυτών. Εμείς ήμασταν πάντα ανοιχτοί και προσπάθησα προηγουμένως να σας πω ότι πολλά πράγματα μπορούν να συνδυαστούν, γιατί λοιπόν όχι και με άλλους τομείς τα κλειστά συστήματα, τα ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό Νομίζω λοιπόν ε, ότι υπάρχουν ε, κλειστά συστήματα, αυτό είναι γνωστό ε, και εδώ υπάρχει πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα καινούργια σκέψη. Κυρία Ράιμα, όσον αφορά τον νόμο περί σπόρων, θεωρώ και νομίζω αυτό το ρώτησε και ο κύριος Χόισλινγκ, εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε την προστασία των καλλιεργητών, τότε πράγματι ε, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε κάποιες ποικιλίε. Και με τον τρόπο αυτό θα ικανοποιήσουμε και εκείνους που ασχαλούνται με τις ε, καλλιέργειες. Το δεύτερο που θέλω να πω, και εδώ ε, παίζουν ρόλο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πράγματι υπάρχει μια ολόκληρη γραφειοκρατία και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί Δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορούμε να το καταργήσουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο εδώ υπάρχει κάτι που μπορούμε να το αναφέρουμε. Όσον αφορά τα ζενιοκτώνα ασθενειών ε, καραντίνας, πράγματι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα ε, και μέχρι τώρα είχαμε προβλήματα και δεν είχαμε κινδύνους που μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Ε, πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα υπόβατρο. Ε, Επιπλέον, κυρία Χόισλινγκ, όσον αφορά την καλλιέργεια και την ανθοκομεία σε τρίτες χώρες, ε, υπάρχει μια λέξη κλειδί, το, το θεμητό εμπόριο, fair trade, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να συμπεριλάβουμε στην παραγωγή και κοινωνικά στοιχεία. Αλλά έχετε δίκιο, αν δούμε λιγάκι τις ε, προδιαγραφές που εφαρμόζουν ε, συνάδελφοί μας ε, και σε μάς την παραγωγή. Πράγματι και εμείς θα θέλαμε αυτά να ισχύουν για εισαγωγές από τρίτες χώρες και για τα οποροκυπευτικά, όχι μόνο για τα καλοπιστικά φυτά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Αν ε, η εισηγήτρια θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Βρήκα πάρα πολύ συγκλονιστική αυτή την ε, συζήτηση. Ευχαριστώ πραγματικά τους ομιλητές για αυτά που μας παρουσίασαν. Η πρόκλησή μου είναι από εδώ και πέρα να λάβω σοβαρά υπόψη μου όλα αυτά στην έκθεσή μου και με μεγάλη χαρά θα συνεργαστώ με τους σκιώδες εισηγητές έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε με την εργασία μας σε κάτι που θα προωθήσει όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα. Αυτά που βρήκα εξαιρετικά σημαντικά και που πρέπει νομίζω να υπογραμμίσουμε είναι πρώτον η έρευνα και ανάπτυξη έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε εφαρμογές χρήσιμες για τους παραγωγούς. Πώς δηλαδή περνάμε από την έρευνα, την επιστημονική έρευνα, στην πράξη. Ένας άλλος τομέας που είναι πολύ σημαντικός για τα Ηνωμένο Βασίλειο είναι πως η καλλιέργεια οποροκυπευτικών θα γίνει μια ελκυστική σταδιοδρομία για νέους. Δεν θα πρέπει αυτός ο τομέας να ελκύει μόνο αυτούς που δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Υπάρχουν πολλές σημαντικές ευκαιρίες προοπτικές για τον τομέα των οποροκυπευτικών στην Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουμε, να το προωθήσουμε, έτσι ώστε ο τομέας αυτός να γίνει ελκυστικός για τους νέους. Τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά προσβλέπω στην επόμενη εβδομάδα θα υποδεχθούμε μία αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στην περιοχή μας, το West Midland. Όλοι όσοι θα είναι παρόντες θα μπορέσουν να δουν στην πράξη κάποια από αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Θα δούμε καλλιέργειες ε, φρούτων, λαχανικών, διακοσμητικών φυτών και πραγματικά νομίζω θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επίσκεψη την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πραγματική πρόκληση. Πολλές φορές ε, δεν ξέρουμε πόσο πλούσιος είναι αυτός ο τομέας. Πόσα πολλά φρούτα, λαχανικά, κατηγορίες ε, φυτών περιέχει ο τομέας αυτός. Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικό τομέα με μεγάλη προστιθέμενη αξία και ξέρουμε ότι πρόκειται για ένα τομέα έντασης εργασίας. Πρόκειται για την παραγωγή της τροφής μας και την παραγωγή από την οποία εξαρτάται η ζωή πολλών μικρών παραγωγών στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας ε, τις δυνατότητες που παρέχουμε για τη διάθεση στην αγορά της παραγωγής αυτών των ε, καλλιεργητών με έμεσο αλλά κυρίως με άμεσο τρόπο στις τοπικές αγορές. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ποιότητα αυτών των προϊόντων γιατί μιλάμε για τη διατροφή μας. Η πρόκληση λοιπόν είναι μεγάλη για όλα αυτά τα προϊόντα και για τα διακοσμητικά φυτά. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που εσύ έχεις αναλάβει αυτόν τον τομέα, εσύ είσαι η συγγήτρια. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας ε, εργασία. Ευχαριστώ άλλη μια φορά την εισηγήτρια τους ομιλητές. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας είναι στις 2 Σεπτεμβρίου. Για τα διάφορα δεν υπάρχει τίποτα. Θα ήθελα λοιπόν να τελειώσουμε τις εργασίες μας. Είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Το Σεπτέμβριο θα πρέπει να έρθετε όλοι δρυμύτεροι. Τα θέματα είναι πολλά. Ραντεβού το Σεπτέμβριο.